Είναι πάντα δύσκολο να προσέρχονται οι συνάδελφοι πέμπτες πρωί, αλλά οι σημαντικότεροι έρχονται. Η σημερινή συνεδρίαση, στη σημερινή συνεδρίαση θα ασχοληθούμε με τα Βαλκάνια. Euh, Και την ΕΠΑ. Ευχαριστώ τον κύριο Κλάμπενχάουρ και τον στρατηγό Δεκερναβόν που θα μας μιλήσουν για τις αποστολές Αλτέα και Πόλου, για το Κωσυφοπέδιο και τη Βοσνία. Δύσκολο να μιλήσει κανείς για τις αποστολές αυτές της ΕΠΑ, γιατί στα Βαλκάνια άρχισαν όλα εκεί, είναι το εργαστήριο της ΕΠΑ και παρά το ότι οι ευρωπαϊκές μας προσπάθειες άρχισαν με βάση μια διαπίστωση αποτυχίας, τώρα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε θετικά αποτελέσματα της Ένωσης σε αυτή την ευρωπαϊκή περιφέρεια. Αρχίζουμε λοιπόν με την αποστολή ΛΕΞ. Όλοι ξέρουμε ότι το κοτσιφοπέδιο παραμένει ένα λεπτό θέμα. Ο Σέρβος Υπουργός Αμήνης είχε έρθει χθε, τον ακούσαμε και δεν θέλουμε σήμερα να επανέλθουμε στα γνωστά για το καθεστώς του κοσυφοπεδίου κτλ. Το Βέλεξ λειτουργεί μέσα σε ένα πολύ ευαίσθητο πολιτικό πλαίσιο λόγω ακριβώς του καθεστώτος του κοσυφοπεδίου αλλά βασίζεται σε μια κοινή δράση, συμφωνία ομόφωνη των 27 χωρών μελών. Δεν υπήρξε καμία διαφωνία. Όσο και να υπάρχουν διαφορετικές τάσεις για το καθεστώς, ως προς την αναγκαιότητα να εφαρμοστεί η αποστολή αυτή. Και εγώ είχα συμμετάσχει στις συζητήσεις για το καθεστώς του Κωσυφοπεδίου και πάντοτε συμφωνούσαμε όποιο και να είναι το καθεστώς να υπάρξει παρέμβαση της Ένωσης. Έτσι λοιπόν το ΕΛΕΞ είναι αποστολή που ποσοτικά τουλάχιστον είναι η πιο σημαντική από όλες αλλά και ποιοτικά διότι ασχολείται με θέματα δικαιοσύνης, τελωνίων και αστυνομίας. Επειδή τα πράγματα παραμένουν δύσκολα, όπως φάνηκε και από την αρχή της εφαρμογής της, οι τοπικοί παράγοντες, Πρίστινα, Βελιγράδη κλπ. έχουν εκφράσει ορισμένες επικρίσεις που μου φαίνονται υπερβολικές και αντιφατικές. Αυτά και για τη δικαστική δράση της αποστολής. Και υπάρχει και μια αντίφαση όταν λέμε ότι υπάρχουν μεν γρήγορα και θεαματικά αποτελέσματα αλλά η δουλειά που γίνεται για το δικαστικό δεν μπορεί να γίνει τόσο γρήγορα αφού απαιτείται εξονυχιστική έρευνα κτλ. Εδώ το ΕΛΕΞ όμως δεν έχει σαν στόχο να, να λέει μόνο θεωρητικά τι συμβαίνει, αλλά να έχει πρακτικά αποτελέσματα. Το θέμα του βορείου τμήματος του Κωσυφοπεδίου είναι μια σημαντική, παραμένει ακόμη προβληματικό. Πώς θα αναπτυχθεί η αποστολή εκεί δηλαδή και με τι χρονοδιάγραμμα Όσοι θέλουν περισσότερο θεαματικά παρά πραγματικά αποτελέσματα βέβαια ε, επικρίνουν την αποστολή αυτή αλλά θα ακούσουμε τώρα τις λεπτομέρειες πρώτα από τον κύριο Κλάμπενχάουερ και μετά από τον στρατηγό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψατε μου καταρχήν να τονίσω ότι για μένα είναι μια μεγάλη τιμή αλλά και μια μεγάλη χαρά να είμαι πάλι ενώπιον της Επιτροπής σας εκπροσωπών της ε, πολιτικές δράσης της ΕΠΑ. Είχαμε συ... συζητήσει μαζί με τον υπεύθυνο των δράσεων στο Αφγανιστάν. Τώρα, σήμερα έχω την χαρά να είμαι μαζί με τον κύριο Κέρμα Μπον για να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί σας σε σχέση με την αποστολή ΕΛΕΞ. Και επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε να μιλήσω στην σεξπυρική γλώσσα. Γιατί, γιατί... Η συνεδρίαση, η σημερινή συνάντηση μάλλον είναι πραγματικά πολύ επίκαιρη γιατί τα γεγονότα τη Κυριακή στη Μητρόβιτσα μας έδειξαν ποιε είναι οι κύριε προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η ULEX του επόμενου μήνε. Εμεί ζητούμε να υπάρξει μια παράταση τη αποστολή μα για δύο χρόνια, αλλά αυτέ οι προκλήσει θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και να είναι το κέντρο των προσπαθειών μα. Τρει προκλήσει βλέπω κύριες προκλήσεις. Καταρχήν, η ULEX έχει περάσει μια μεταποιητική περίοδο, μια περίοδο μεταμορφώσεων, σε ό,τι αφορά τις δημόσιες έρευνες και τις κατοίκων έρευνες, σε ό,τι αφορά θέματα καταγγελιών διαφθορά στο δημόσιο τομέα, που έχουν δημιουργήσει και μια ατμόσφαιρα στην κοινή γνώμη. Έχουμε επομένως δημιουργήσει τη βάση για μια σημαντική βελτίωση και ενίσχυση του κράτους δικαίου στο Κωσυφοπέδιο. Όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, η αντιμετώπιση αυτών των ερευνών θα, θα, θα χρειαστεί χρόνο και υποστήριξη όχι μόνο από εσά και από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης <clears throat> αλλά και από τους διεθνείς εταίρους μας. Εμείς βασιζόμαστε στον προνομιακό διάλογο που έχετε αναπτύξει με το Κωσυφοπαίδιο για να στείλετε ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ του κράτους δικαίου και του ρόλου της ULEX. Η πρόοδός μας συνεχίζεται σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της διαφθοράς και του οργανωμένου κλίματος. Η αποστολή μας λειτουργεί όχι μόνο στην Πριστίνα, αλλά και σε όλο το Κωσυφοπαίδιο. Φυσικά η κατάσταση στο βόρειο μέρος του Κωσυφοπαιδίου και αυτό είναι το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να σταθώ έχει πολλά προβλήματα και σημαντικές προκλήσεις. Η σημαντική επιχειρησιακή πρόοδος στον τομέα αυτό θα εξαρτηθεί από μια κοινή αντίληψη όλων των εμπλεκομένων για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να υπάρξει πρόοδο στα θέματα του κοσμοπεδίου. Διαμέσως η αποστολή μας θα συνεχίσει να δρά βήμα με βήμα για να μπορέσει να έχει μια μεγαλύτερη παρουσία στο, βο... στο βορρά του κοσμοπεδίου για να αυξηθούν και οι ενέργειες εφαρμογής του νόμου και λειτουργίας των δικαστικών αρχών. Μας ενδιαφέρει να μπορέσουμε να επανεσωματώσουμε τους Σέρβους δικαστικούς στο Κωσυφοπαίδιο. Σας είπα ότι η πρόοδος σε πολλούς τομείς μπορεί να είναι δύσκολη για τις επόμενες εβδομάδε, αλλά εμείς θα εξακολουθήσουμε να πιέσουμε για να επιτευχθεί κάποια πρόοδος και πιστεύουμε ότι θα ανοίξουν και πάλι τα δικαστήρια στην περιοχή αυτή. Μια άλλη προϋπόθεση βέβαια είναι να υπάρξει σταθερότητα στο βορρά του κοσκοπεδίου και να μπορέσει να λειτουργήσει αποτρεπτικά η παρουσία δύναμη της ULEX. Εν παραλίλω, θα συνεχίσουμε και αυτήν την η τρίτη μου παρατήρηση, να ενισχύουμε την επαγγελματικότητα των θεσμών του κοσκοπεδίου για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και την βιωσιμότητα των προσπαθειών μας και εν καιρό να, επιτρέψουμε, να επιτρέψουμε μια βαθμία μετάβαση και μεταφορά εξουσιών επί τη βάση αντικειμενικών κριτηριών και benchmarks. Αυτή είναι και η βάση της ε, εταιρική μας σχέσης με τις αρχές του Κωσυφοπεδίου και η παράταση της, οδηγίας. της ε, εντολής τη Αγιούλεξ πρέπει να ειδωθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Είναι φυσιολογικό φυσικά μέσα σε αυτό το πλαίσιο να τονίζουμε ότι πρέπει οι αρχές του κοσμοπεδίου να αναλάβουν μεγαλύτερο ρόλο σε ό,τι αφορά το κράτο δικαίου και την εφαρμογή του. Αυτά ήθελα να σας πω λοιπόν εισαγωγικά και θα ήθελα τώρα να σα ξαναδώσω το λόγο. Ευχαριστούμε κύριε Κλόμπεν Χάουερ, ο κύριο Κάμε Μπον. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω καταρχάς ότι είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ ενώπιόν σας για να σας ενημερώσω για την κατάσταση της αποστολής Γιούλεξ στο Κοσφοπέδιο. Θα ήθελα καταρχάς να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είχα έρθει εδώ στις 27 Απριλίου. Αλλά Τελευταία στιγμή χρειάστηκε να κυρώσω το ταξίδι μου στις Βρυξέλλες λόγω σημαντικών εξελίξεων στο κοσφοπέδιο που απέτησαν την παρουσία μου στην Πριστίνα. Μιλάω για, τις, για την κατάσταση στο Υπουργείο Μεταφοράς και Επικοινωνιών. Ε, ήμουνα με την κυρία Γιουνέσο στην Πρίστινα Καταλαβαίνετε, ελπίζω, την ε, ανάγκη ε, να οργανώσουμε την ε, συνάντηση εκείνη της 27 Απριλίου αργότερα. Θα σας κάνω όμως σήμερα μια παρουσίαση που αποτελείται από τρία μέρη. Θα ξεκινήσουμε με μια σύντομη εισαγωγή των βασικών χαρακτηριστικών της αποστολής, εν συνεχεία θα σας μιλήσω για τις, ε, τα, της, ε, τα κύρια επιτεύγματα της αποστολής και τέλος θα σας μιλήσω για τις προκλήσεις της αποστολής. Να σας μιλήσω για τα βασικά καταρχάς χαρακτηριστικά της αποστολής. Η Ulex, όπως τα ξέρετε, είναι η μεγαλύτερη αποστολή ΕΠΑ με προσωπικό 1.717 ανθρώπους και 1097 ντόπιου. Τα άτομα του προσωπικού είναι πολίτες και των 27 ε, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, της ε, Ρωσίας, ε, Νορβηγίας και Τουρκίας. Ο προϋπολογισμός είναι 155 εκατομμύρια ευρώ. Και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό ε, στο συνολικό προπολογισμό της ΕΠΑ. Είναι η πρώτη αποστολή της ΕΠΑ με μια εκτελεστική εντολή που είναι πολύ σημαντικό. Αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι ο πυρήνας των δραστηριοτήτων της αποστολής είναι το monitoring, η αξιολόγηση και η συμβουλή των αρχών του πεδίου. Υπάρχει λογοδοσία από μέρους μας και αξιοπιστία. Οι αρχές του κοσμοπεδίου είναι αυτές που έχουν την πρωτοκαθεδρία. Θα πρέπει να πετύχουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο και εμείς είμαστε εκεί απλώς να τους βοηθήσουμε. Όταν συναντήθηκα με τον Πρωθυπουργό, τόνισα ότι οι αρχές του κοσμοπαιδείου θα πρέπει να έχουν το προβάδισμα για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Συμφωνούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια έντονη εταιρική σχέση μεταξύ μας. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Γιούλεξ είναι τεχνική αποστολή, δεν είναι πολιτική αποστολή. Η εντολή της είναι σαφής, αφορά το κράτος δικαίου και όχι το καθεστώς του κοσφοπεδίου, κύριε Πρόεδρε. Περιτώ να σας υπενθυμίσω ότι η κοινή δράση της Ιούλεξ υιοθετήθηκε και από τα 27 κράτη-μέλη και εκείνα που δεν αναγνωρίζουν την ανακρατησία του κοσμοπεδίου. Η εντολή λοιπόν της αποστολής είναι σαφής και εκτελείται μέσα στα μέσα και τις δυνατότητε που έχουμε ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τελευταίο βασικό χαρακτηριστικό της αποστολής που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι ενσωματώνεται, ότι έχει μια ολοκληρωμένη φύση. Αστυνομία, ε, δικαιοσύνη και τελωνία είναι οι τρεις τομείς και ο συντονισμός αυτών των ε, δραστηριοτήτων είναι πολύ σημαντικό για την επιτυχία της αποστολής. Είναι ολοκληρωμένη λοιπόν αποστολή. Δεν είναι εύκολο καθήκον αυτό, ε, γιατί το κοσμοπέδιο είναι ένα δύσκολο περιβάλλον οι, τα μέλη του προσωπικού έχουν τελείως διαφορετική προέλευση, πολιτισμό, θρησκεία κτλ. Ο συντονισμός μεταξύ της δικαιοσύνης και της αστυνομίας επιτόπου ε, δεν είναι καθόλου εύκολο. Η συνιστόσα της αστυνομίας είναι η πιο μεγάλη. Ε, συμπεριλαμβάνει το... τα τμήματα της αστυνομίας, το ειδικό τμήμα της αστυνομίας, τις ειδικέ αστυνομικές δυνάμεις. Το δεύτερο είναι της δικαιοσύνης με 18 από τις 25 και 66 από 71 δικαστές. Ζητάμε συνέχεια από τα κράτη-μέλη να μας δώσουν δικαστές και εισαγγελείς, αλλά δεν έχουμε αρκετό προσωπικό ακόμα θα ξαναμιλήσω για αυτό το θέμα στο τελευταίο τμήμα της παρουσίασής μου. Υπάρχει πλήρως, πλήρης σεβασμός ανεξαρτησίας των δικαστών και της αυτονομίας των εισαγγελέων. Αυτές οι αρχές είναι θεμελιώδεις, παρότι το περιβάλλον εργασίας σε μια αποστολή με μια περίπλοκη εντολή όπως αυτή στο Κοσμοπέδιο είναι τελείως διαφορετικό από το σύνηθες εργασιακό περιβάλλον αυτών των δικαστών και εισαγγελέων. Ε, και τα τελωνία. Η τελωνιακή συνιστόσα είναι η μικρότερη, αλλά αυξάνεται γιατί μπορεί να χρειαστεί να εκτελέσει στο βόρειο κοσμοπέδιο και επιπλέον καθήκοντα. Θα επανέλθω και σε αυτό το σημείο αργότερα. Επομένως, θα ήθελα να δούμε τώρα κάποια από τα επιτεύγματα της αποστολής. Καταρχάς, θα ήθελα να ξεκινήσω τονίζοντας ε, τι έχει κάνει η Γιούλεξ συνολικά στο κοσφοπέδιο. Ε, στη φάση του σχεδιασμού δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα είχαμε τέτοιες ε, επιτυχίες. Μιλάω για το ψήφισμα του ΟΗΕ και τις συζητήσεις της Τρόικα στο τέλη του 2007, καθώς και τις προπασκευαστικές συνομιλίες στην Ουάσιγκτον. Μετά την δήλωση το Φεβρουάριο του 2008 της ανεξαρτησίας του Κοσφοπέδιου, δύο τελωνιακοί στο Κοσφοπέδιο σκοτώθηκαν και, και στη Μητροβίτσα α, υπήρξε λαϊλασία των, ενός δικαστηρίου. Παρά την ε, ένταση αυτή λοιπόν και τις φοβερές ε, τεχνικές δυσκολίες και, τις, και οι τρεις ε, συνιστός της ULEX ε, αναπτύχθηκαν με επιτυχία στις 9 ε, Δεκεμβρίου 2008. Ξεκίνησε τότε η αποστολή αυτό, έγινε σε όλο το κοσμοπέδιο. Η συνιστόσα της α, ε, δικαιοσύνης και του τελωνίου στην αρχή και εν συνεχεία οι υπόλοιποι συνιστώσεις. Όλα αυτά συνέβησαν χωρίς, ε, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το προσωπικό της ε, Γιούλεξ ε, πήγε, τα πήγε θαυμάσια. Και θα να ευχαριστήσω όλους όσους συνεισέφεραν στην επιτυχία αυτού που θεωρούσαμε ανέφικτη αποστολή. Mission impossible. Ε, το Βόρειο Κοσμοπέδιο είχε γίνει ένα είδος περιοχής duty free. Γι' αυτό με μεγάλη χαρά, όταν διάβασα την ακόλουθη αρχή ε, δήλωση στα ΜΜΕ, ότι ο Γενικός Διευθυντής του, των Τελωνίων στις 23 Μαρτίου του 2010 ανέφερε ότι πέρυσι τα πήγαμε πολύ καλύτερα από τις προηγούμενες χρονιές καταφέραμε να καταπολεμήσουμε το κρίμα, το έγκλημα και το λαθρεμπόριο. Και μειώθηκε το έγκλημα. Το λαθρεμπόριο, συγγνώμη, μειώθηκε κατά 80%. Οι τοπικοί εγκληματίες προσπάθησαν να εμποδίσουν την Γιούλεξ να δραστηριοποιηθεί με οδοφράγματα προσπάθησαν αλλά απέτυχαν. Και η Γιούλεξ λοιπόν ε, παρέμεινε παρούσα. Αυτό έγινε χάρη στην συνεργασία με την K4 που μας υποστήριξε όταν το χρειαστήκαμε. Θα ήθελα να τονίσω ότι η συνεργασία με την K4 σε όλα τα επίπεδα ε, δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Είμαι σε συνεχή επαφή με την K4 και το στρατιωτικό μου παρελθόν με βοήθησε για να καταλάβω τι θα μπορούσα και τι δεν θα μπορούσα να ζητήσω από την K4. Επίσης είχα προηγούμενες διαμονές στο κοσφοπέδιο που με βοήθησαν να προσαρμοστώ και να καταλάβω το περίπλοκο αυτό περιβάλλον. Τώρα, ένα άλλο σημαντικό επίτευγμα είναι το γεγονό ότι πριν από ένα χρόνο οι Σέρβοι και οι Αλβανοί άρχισαν να ξαναχτίζουν τα σπίτια τους σε εθνικά μεικτές περιοχές του βορείου Κωσυφοπεδίου. Οι οικίες τους είχαν καταστραφεί κατά τη διάρκεια του πολέμου και είχαν μείνει ακατοίκητα για πάνω από 10 χρόνια. Υπήρξε αντίδραση από την πλευρά των Σέρβων για την ανοικοδόμηση αυτή και ξεκίνησε εθνοτική βία. Αυτό ήταν μια πραγματική δοκιμασία για την ULEX. Αλλά και η αστυνομία του Κοσφοπέδιου επελήφθη του θέματος αυτού. Μπορέσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση με επιτυχή τρόπο. Η K4 ήταν έτοιμη, υπήρξε πλήρης συντονισμός με τη ULEX, αλλά δεν χρειάστηκε να παρέμβει η ισχυρή θέληση της ε, EULEX να χρησιμοποιήσει στρατιωτική της δύναμη με αναλογικό τρόπο σε αυτό το πολύπλοκο πλαίσιο χωρίς απώλεια ζώων έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο και συνέβαλε τα μάλα για να υπήρξε <clears throat> μια ε, παράταση της ε, παρουσίας της KFOR στο Κωσυφοπέδιο και αυτό ενίσχυσε και την ικανότητα επιβολής του νόμου στην περιοχή. Θέλω επίσης να σας υπενθυμίσω το πόσα πράγματα εκκρεμούν μετά από τη θητεία της Ιουν και το γεγονός ότι είναι πολύ αποδυναμωμένη δικαστική εξουσία στην περιοχή. Η δικαστική μας συνιστόσα πήρε πρόσβαση στα δικαστικά αρχεία μόνο πρόσφατα. Η πρόσβαση σε απαραίτητο χώρο γραφείων για την μονάδα αυτή της UNMIC οδήγησε σε πολλά προβλήματα ε, και καθυστέρησε προτού να υπάρξει ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Για μας είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρξει μια καλύτερη και πιο οικοδομητική κατανόηση της κατάστασης. Δεν θα σας κάνω να νιώσετε κόποση με όλες τις περιπτώσεις που θα μπορούσα να σας αναφέρω σε αυτή την περίπτωση του κοσμοπεδίου. Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις διαφθοράς, ε, οργανωμένου εγκλήματος, τρομοκρατίας, εγκλήματων πολέμου, εθνοτικής βίας κτλ. Εμείς όμως είμαστε παρόντες σε όλα τα δικαστήρια και σε όλα τα δικαστικά επίπεδα. Στο τομέα του οργανωμένου εγκλήματος, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, θέλω να σας φέρω, φέρω στην προσοχή σας το γεγονός ότι, το γεγονός ότι πρόσφατα οι σερβικές δικαστικές αρχές προσκάλεσαν μάρτυρες να καταθέσουν στη Σερβία ενώπιον ενός δικαστή ανακριτή. Οι Κωσοβάροι δεν δέχτηκαν αυτή την αίτηση και υπήρξαν και δύο επεισόδια κατά των ε, μαρτύρων. Αυτό όμως είναι ένα σημαντικό στοιχείο συνεργασίας μεταξύ Βελιγραδίου και Πριστίνες. Η Γιουλέξ έχει παίξει ένα μεγάλο ρόλο μέχρι στιγμή στο να διευκολύνει τη διαδικασία αυτής της συνεργασίας και βάσει της άποψης ορισμένων εμπειρογνωμών η συνεργασία στα θέματα αυτά είναι μια θετική, ίσως η πιο θετική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Επίσης, ανακαλύψαμε ένα, ε, ένα κοινό τάφο στην περιοχή της Άσκα. Και αυτό έγινε με τη συνεργασία και της Ιουλέξης και τα θέματα αυτά και των σερβικών αρχών. Εμείς έχουμε χρησιμοποιήσει και την ικανότητα συνεννόηση με το Βελιγράδι πολλές φορές και εγώ πήγα δύο φορές στο Βελιγράδι. Πήγα στην, στα Σκόπια, στην Κόρτζα και στα Τύρανα ω τμήμα της ε, δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίσουμε ζητήματα όπως αυτά του οργανωμένου εγκλήματος. Η Γιούλεξ έχει ένα περιφερειακό γραφείο στο Βελιγράδι και πηγαίνουμε τακτικά εκεί για τεχνικές ε, συναντήσεις με τον Υπουργό Δικαιοσύνη και άλλους αξιωματούχους Εργαζόμαστε σε στενή συνεργασία με τον Πίτερ Φρόνσεν που είναι ο προσωπικός εκπρόσωπος του, της υψηλής εκπροσώπου στο Βελιγράδι. Έχουμε υπογράψει ένα πολιτικό πρωτόκολλο με το Βελιγράδι που μας επέτρεψε να έχουμε επίσημα ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα. Και η αποστολή μας εργάζεται για να πετύχει αντίστοιχες τεχνικές ρυθμίσεις για το θέμα των τελωνιακών ελέγχων η Ulex αντιμετωπίζει τώρα τον πυρήνα του, της εντολής της πολέμηση οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς. Η έρευνε που έγινε στο Υπουργείο Επικοινωνιών και Μεταφορών είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, ένα αυτό παράδειγμα αυτών των προσπαθειών. Βρισκόμαστε μόνο στην αρχή. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι έχουν βοηθήσει σε τοπικό πολιτικό επίπεδο και για την υποστήριξη που μας έδωσαν όταν έπρεπε να ληφθούν δύσκολες πολιτικές αποφάσεις. Χαίρομαι που η κυβέρνηση του Κοσμοπεδίου το Μάρτιο θέσπισε μια ομάδα δράσης κατά της διαφθοράς μέσα στο Γραφείο Ειδικών Ερευνών και Διώξεων με πέντε ε, ανακριτές από το Κόσοβο και τρεις από, από, από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητήσαμε να υπάρξει μια αξιολόγηση από τη δική του πλευρά για να δούμε πώς μπορούμε στο μέλλον να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα αυτής της δύναμη και στη συνέχεια ο Πρωθυπουργό και εγώ πήγαμε στην μονάδα αυτή και τονίσαμε προ τα μέσα ενημέρωση τη μεγάλη σημασία που αποδίδουμε στον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματο και της διαφθοράς αλλά μέσα, στα μέσα σε ένα πνεύμα συνεργασίες. Η να παίρνει αυτή τη συνεργασία πολύ σοβαρά και θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν γιατί χάρη σε αυτήν μπορούμε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή. Είναι ένα από πολλά παραδείγματα της θαυμάσιας συνεργασίας που έχουμε με τις τοπικές αρχές. Σε ό,τι αφορά τους ε, ομολόγους μας, επίσης θα ήθελα να τονίσω την σημασία της συνεργασίας μας με όλους τους εμπλεκόμενους στο Κοσμοπέδιο. Ο Πρωθυπουργός με τον οποίο έχω τακτική επαφή έχει πάντα τονίσει το ενδιαφέρον που έχει για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει δείξει μεγάλη πολιτική οριμότητα όταν η κυβέρνησή του αντιμετώπισε τις έρευνες σε ένα από τα Υπουργεία τους. Το Συμβούλιο Συντονισμού, όπου συμμετέχω μαζί με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, συναντάται κάθε έξι εβδομάδες, συναντάται για να συζητήσει στρατηγικά θέματα με παρουσία του Υπουργείου Εσωτερικών Δικαιοσύνης και Οικονομικών. Γίνεται λοιπόν αυτή η επίσης συνάντηση σε άτυπο επίπεδο μια φορά την εβδομάδα. Θέλουμε επίσης να εξασφαλίσουμε και την επαφή με την κοινωνία των πολιτών του Κωσυφοπεδίου. Σε σχέση με το κατά πόσο είναι υπόλογη σε πολιτικό επίπεδο η αποστολή μας, <clears throat> θέλω να τονίσω ότι η πρώτη συνεδρίαση του πάνελ για τα ανθρώπινα δικαιώματα έλαβε χώρα. Αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα γιατί χρειάστηκε η UNMIC προσπάθειες μιας δεκαετίας για να επιτύχει κάτι τέτοιο. Αλλά πρέπει να εστιάσουμε την προσπάθειά μας στο βόρειο τμήμα του Κοσμοπεδίου. Αυξάνουμε την παρουσία μας στο βόρειο τμήμα του Κοσμοπεδίου μαζί με τους άλλους εταίρους μας στον του Βασιλείο. Βασιλείου. 20 Μαρτίου μαζί με τον Ιταλό πρεσβευτή και την Κομισιόν διοργανώσαμε μια πρώτη ε, τοπική διάσκεψη τύπου στη Μητρόβιτσα και αυτό δείχνει την παρουσία μας. Είμαστε έτοιμοι να αυξήσουμε λοιπόν την ορατότητά μας στην περιοχή αυτή. Η αστυνομία και οι τελωνιακές αρχές έχουν αυξήσει τις δράσεις τους για να καταπολεμήσουν τις παράνομες ενέργειες και το οργανωμένο έγκλημα. Η έλευση των 15 τελωνιακών οι οποίοι είχαν προσληφθεί μας επέτρεψε να τροποποιήσουμε την ε, την ε, δράση μας εκεί και να βελτιώσουμε και την ε, αποτελεσματικότητά μας. Και σιγά σιγά προχωρούμε προς πλήρη τελωνιακό έλεγχο. Συντονίζουμε τις προσπάθειές μας με τις ΗΠΑ, με την ε, Κομισιόν και με άλλους εμπλεκόμενους. Υπάρχουν κάποιες πτυχές αυτού του θέματος, όπως η κατανομή φορολογικών εσόδων, που φυσικά έχουν πολιτικό χαρακτήρα και εκφεύγουν τις εντολίες μας. Η αστυνομική αρχή, οι αστυνομικές αρχές επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουν και την πλήρη στελέχωση όλων των αστυνομικών σταθμών στο βόρειο τμήμα του Κωσυφοπεδίου. Έχει υπάρξει λοιπόν μεγάλη ευκαμψία και ικανότητα να διατηρηθεί η δικαστική παρουσία στη Μητρόβιτσα παρά τις καταστροφές τμήματος αυτού του κτηρίου κατά τη διάρκεια του σεισμού της 10 Μαρτίου. Η συνέχεια λοιπόν στο δικαστικό τομέα, στο βόρειο τμήμα του Κωσυφοπεδίου, είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα προς όλες τις κοινότητες. Θέλω να εξάρω το σημαντικό έργο των διοικητικών αρχών που έπαιξαν κεφαλαιόδη ρόλο για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια και τη συνεχιζόμενη πρόσβαση στο κτίριο αυτό. Όλα αυτά είναι μικρά βηματάκια, αλλά προς τη σωστή κατεύθυνση. Ξεκινήσαμε με προσωπικό της ε, ULEX, μετά προσθέθηκε προσωπικό από το Κοσφοπέδιο και έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια να εξασφαλίσουμε την επανενσωμάτωση δύο Κωσοβοαλβανών και δύο Σέρβων δικαστικών. Σιγά σιγά θα εξασφαλίσουμε την πλήρη ομαλοποίηση του κράτους δικαίου στο Βόρειο Κωσφοπέδιο. Πρέπει όμως να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορέσει να εδρεωθεί αυτή η κατάσταση πρωτού προχωρήσουμε προς τα επόμενα βήματα γιατί εξακολουθεί να είναι δύσκολη κατάσταση η πολιτική μας ήταν επιτυχής και δεν χρειαστήκαμε σε καμία περίπτωση να υποχωρήσουμε. Θέλουμε να συνεχίσουμε λοιπόν τις δράσεις μας. Υπάρχει και το θέμα της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς των Σέρβων στο Κοσφοπέδιο. Είμαστε σε επαφή με την, τους της Ορθόδοξης Εκκλησίας ε, των Σέρβων στο Κοσφοπέδιο και χαίρομαι για αυτές τις επαφές στον Καζί Μεστάν στις 18 Μαρτίου υπήρξε μια τέτοια συνάντηση όπου η ULEX ε, συντόνισε τις δράσεις της αστυνομίας του Κωσικοπεδίου. Εγώ μαζί με τον ε, Υπουργό Εσωτερικών επισκέφθηκα την περιοχή στις 20 Μαΐου και ήμουν πολύ ικανοποιημένο με τα πορίσματα αυτά. Είμαι σε στενή επαρχή με τον Έλληνα πρεσβευτή, ο οποίος παίζει διευκολυντικό ρόλο επίσης για τις δράσεις αυτές. η επιδιώκωση των εκκλησιών είναι ένα επίσης από τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν με τους ε, συνομιλητέ μας από την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών και όπως τόνισα η σχέση μας με την ΚΕΙΦΟΡ είναι η καλύτερη δυνατή και αυτό αναφέρθηκε και στη σύνοδο του, Μα... του Μαΐου του ΝΑΤΟ. Έρχομαι τώρα στο τρίτο τμήμα για τις προκλήσεις για τις προκλήσεις. Πριν όμως θα ήθελα να σας αναφέρω τις διοικητικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Έχουμε ακόμη τέτοιες ελλείψεις και δυστυχώς οι ισχύουσες διαδικασίες δεν μπορούν να το λύσουν. Ή τουλάχιστον σύντομα δεν μπορούν να το λύσουν. Το 2007 είχε ζητηθεί η γρήγορη ανάπτυξη 2.000 ανδρών προσωπικού και χιλίων τοπικών. Αλλά αυτό δεν μπόρεσε να γίνει όπως προβλεπόταν από το σχέδιο γιατί οι διεθνείς πολιτικές δυσκολίες μας δημιούργησαν τεράστια προβλήματα. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω μία συγκεντρωτική διαχείριση του υλικού που διαθέτουμε. Γιατί έτσι θα αυξηθεί η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητά μας. Πολλά θα μπορούσαμε να κερδίσουμε αν γινόταν μια σωστή μελέτη της χρήσης του υλικού που διαθέτουμε. Σας έχω ήδη πει ότι η αποστολή χρειάζεται περισσότερο προσωπικό. Θα σας ήμουν ευγνώμων αν μπορούσατε να πιέσετε τις πρωτεύουσές σας για να αυξηθεί. Αυτό είναι πρόβλημα που υπάρχει από την αρχή. Πρέπει τα μέλη της αποστολής όταν επιστρέφουν από τα, στις χώρες τους από τα καθήκοντά τους εκεί να κάνουν και μία αξιολόγηση. Και αυτό θα μπορούσε να γίνει καλύτερα μέσω συγκεντρωτικής διαχείρισης και του προσωπικού. Έτσι θα ήταν καλύτερη και ευθυνότερη η διαχείριση και θα μπορούσαμε να ελέγξουμε καλύτερα και την επαγγελματική εμπειρία που διαθέτει το προσωπικό αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν για τις προσπάθειές της σχετικά, αλλά η οικονομική διαχείριση της θα έπρεπε, αν είναι δυνατόν, να αλλάξει έτσι ώστε οι αλλαγές του προσωπικού να γίνονται γνωστές εγκαίρως για να πληροφορείται και το προσωπικό για τις αλλαγές αυτές. Τέλος, το κράτος δικαίου που θέλουμε να δημιουργήσουμε στο κοσυφοπέδιο θέλουμε να συμφωνεί με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Σκοπός μας δεν είναι να διαχειριστούμε εμείς το κοσυφοπέδιο, Βέβαια ορισμένα από τα προγράμματά μας θα έχουν πολιτικές επιπτώσεις αλλά η ΕΛΕΞ δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα. Τα πολιτικά, με τα πολιτικά ασχολούνται άλλοι. Εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε την ενότητα της αποστολής και κυρίως να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία των δικαστικών. Αυτά είναι ευρωπαϊκές αξίες. Θέλουμε να διατηρήσουμε την αρχική ορεμή της αποστολής. Ο βοράς του Κωσυφοπεδίου είναι ιδιαίτερο πρόβλημα και θα πάρουμε μαθήματα από τις επιτυχίες που σημειώσαμε στο Νότο. Είμαστε ευγνώμονες για τη βοήθεια που μας δίνει η Βρυξέλλες, ιδίω στο πρόσωπο της κυρίας Άσιτον. Σας κατευχαριστώ για την προσοχή σας και με μεγάλη ειδονή θα απαντούσα σε τυχόν ερωτήσεις. Euh, σας ευχαριστώ και τους δύο για τις εξαντλητικές σας παρουσιάσεις. Θα ακούσουμε τώρα τις αντιδράσεις των συναδέλφων. Συλλογικά σας ζητούμε συγγνώμη για τη συνεδρία της 27ης Απριλίου που χρειάστηκε να αναβληθεί αλλά ήταν απαραίτητο και βλέπετε και εσείς τώρα, ε, καταλαβαίνετε και εσείς γιατί, γιατί χρειαζόταν στην Πρίστινα να γίνουν διάφορα πράγματα. Δεν ξέχασα να σας πω στην παρουσίαση ποιο είναι το στρατιωτικό σας παρελθόν, ήσασταν μέλος και της ΚΦΟΡ από πολλά χρόνια και έρχομαι έτσι σε ένα ερώτημα ή μια απορία που μας ταλανίζει εδώ πέρα πώς συνδέονται οι αποστολές ΕΠΑ με τις αποστολές του ΝΑΤΟ. Στο Αφγανιστάν και το Κωσυφοπέδιο η απουσία συμφωνίας μεταξύ Ένωσης και ΝΑΤΟ θέτει προβλήματα τεχνικά επιτόπου. Πιο φανερά, πιο θεαματικά στο Αφγανιστάν παρά στο Κωσυφοπέδιο, αλλά και εσείς ως επικεφαλής της ΚΦΟΡ Θα μπορούσατε να μας πείτε ποια είναι ακριβώς αυτά τα προβλήματα διασύνδεσης, ποιος κάνει τι, ιδίω για τη διατήρηση της τάξης και ποια είναι η ακριβή σύνδεση μεταξύ της κοσυφοπεδικής αστυνομίας της ΕΛΕΞ και του ΝΑΤΟ. Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω κάτι πιο πολιτικό τι επιπτώσεις θα έχει η εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας ως προς τις εξωτερικές δράσεις στην ορατή παρουσία της Ένωσης στο κοτσιφοπέδιο γιατί και εγώ όταν πήγα εκεί διαπίστωσα πέντε τουλάχιστον ευρωπαϊκές σημαίες σε πέντε διαφορετικά κτίρια ευρωπαϊκών κρατών μάλλον πράγμα το οποίο ε, δεν διευκολύνει την αξιοπιστία της αποστολής ούτε τη γνώση του ποιος κάνει ακριβώς τι. Εσείς ακριβώς τι κάνετε και πώς τα συνδέετε όλα αυτά με τη δράση των υπολείπων για να υπάρχει μεγαλύτερη ορατότης και συνέπεια. Αυτά ήθελα να σας πω και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Λούνατσεκ, εισηγήτρια επί του Κωσυφοπεδίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας κύριε Ντεκερμαμπό και εγώ δέχομαι τη συγγνώμη σας. Καταλαβαίνω την κατάσταση γιατί και εγώ έχω πάει στην Πρίστινα και ξέρω ποια είναι η κατάσταση. Παρότι οι διάφοροι συνάδελφοι απογοητεύτηκαν ε, που δεν ήσασταν εδώ στις 27, εγώ ήμουν στην Πρίστινα στις 28 και κατάλαβα γιατί δεν ήρθατε εδώ στις 27. Αυτά. Τώρα θέλω να ξεκινήσω την παρέμβασή μου με κάποια συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνει η Γιούλεξ. Ξεκινάνε ανακρίσεις και έρευνες. Έγιναν οι έρευνες στο Υπουργείο Μεταφορών, ακόμη και στα γραφεία του Υπουργού και στο σπίτι του. Η Γιούλεξ είχε πει ότι θέλει να προχωρήσει και θέλει να ερευνήσει και τα μεγάλα ψάρια της διαφθοράς. Και τελικά τέλη Απριλίου κατάλαβα από τις επαφές που είχαμε ανθρώπους στο δρόμο, στο αεροδρόμιο, στα εστιατόρια. Ο κόσμος έχει αυτή την αίσθηση ότι κάτι κάνει η Γιούλεξ. Έχει λοιπόν ο κόσμος πραγματικές προσδοκίες από τη Γιούλεξ. Να μην παίξει το ρόλο του χωροφύλακα μόνο, αλλά να προχωρήσει και με τη διαφθορά, να κάνει κάτι για τη διαφθορά. Τρεις φορές έχω πάει στο Κοσφοπέδιο και οι Κοσοβάροι έχουν πραγματικές προσδοκίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τη Γιούλεξ, γιατί πιστεύουν ότι το δικό του σύστημα δεν είναι αρκετά δυνατό για να τους βοηθήσει. Η διαφθορά υπάρχει στην καθημερινή ζωή και θέλουν οι θύνοντες, ακόμη και αν βρίσκονται ψηλά, να διωχθούν, αν είναι υπεύθυνοι διαφθοράς ή οργανωμένου εγκλήματο. Επομένω αυτέ οι έρευνες είναι πολύ σημαντικές για τους πολίτες, για την κυβέρνηση, αλλά και για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κοσμοπέδιο. Όταν ε, υπήρξε η δήλωση της ανεξαρτησίας, όταν δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα, επειδή όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνώρισαν το καθεστώ ανεξαρτησία του Κωσυφοπεδίου. δημιουργήθηκε αυτή η ένταση με το Κωσυφοπεδίο. Γι' αυτό χρειάζεται αυτή η αξιοπιστία. Και είναι σημαντικό ότι και τα 27 κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση σα έδωσαν την εντολή να κάνετε, να προχωρήσετε με την αποστολή. Ε, χαίρομαι για όλα αυτά που κάνουν οι δικαστές, οι εισαγγελείς. Αυτό που θέλουν είναι να προχωρήσουν ως το τέλος. Τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξαν πιέσεις από κάποιους κύκλους. Εν μέρη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από κυβερνήσεις κρατών μελών που φοβούνται ότι αν συνεχιστεί αυτή η οδός μπορεί να υπάρξει πρόβλημα σταθερότητας στο κοσμοπέδιο. Εγώ δεν πιστεύω κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι τώρα πια, όπως φάνηκε και τα τελευταία δύο χρόνια, έχει μπει σε μία φάση ομαλοποίησης. Δεν υπάρχουν δύο επεισόδια, υπάρχει σταθερότητα. Επομένως είναι σημαντικό απλώς να είμαστε εκεί και να υποστηρίξουμε το κράτος δικαίου. Να φτάσουν αυτές οι ανακρίσεις μέχρι το τέλος και αυτό τι σημαίνει. Ακόμη και να κατηγορηθούν και να παραπευθούν στη δικαιοσύνη υπουργοί. Αν χρειάζεται, έτσι. Αν δεν είναι υπεύθυνοι, φυσικά θα αθωωθούν. Αλλά δεν πρέπει να σταματήσουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε μέχρι του ηθήνοντε. Σα ευχαριστώ λοιπόν για όλα όσα κάνατε, για το πώ χειρίζεστε την κατάσταση. Ξέρω είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και για εσά και δεν έχει τελειώσει ακόμα. Αλλά είναι σημαντικό να φτάσουμε μέχρι το κόκαλο, μέχρι του ηθήνοντε. Να ξεκαθαριστεί η κατάσταση. Κοιτάξτε, η στάση πρέπει να είναι αμερόληπτη της Γιούλεξ. Ε, να στραφούμε παντού, όχι προς συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα, όχι προς το πολιτικό κόμμα, ας πούμε, του Πρωθυπουργού. Οποιοδήποτε, όπου και αν βρίσκεται, αν ε, συμμετείχε σε οργανωμένο έγκλημα, αν είναι υπόλογος διαφθοράς, να διωχθεί, να δικαστεί. Είναι σημαντικό αυτό για τη χώρα. Ε, ένα άλλο πρόβλημα που αναφέρατε είναι ότι δεν έχετε επαρκές ε, προσωπικό. Έχετε περίπου 50 ε, δικαστές και εισαγγελείς, 1.500 αστυνομικούς και περίπου καμιά τριανταριά τελωνιακούς. Κάτι άλλο που το έχω γράψει και στην έκθεσή μου. Είναι σημαντικό να αποσπάσουν περισσότερους δικαστές και εισαγγελείς Είπατε ότι εμείς πρέπει να μιλήσουμε στις κυβερνήσεις μας για να βοηθήσουμε. Αλλά τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να πείσουμε τις κυβερνήσεις μας να στείλουν περισσότερους δικαστές και εισαγγελείς. Γιατί έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν υπερβολικά πολλοί αστυνομικοί και ξέρουμε ότι η αστυνομία του Κωσυφοπεδίου ε, κάνει πολύ καλή δουλειά. Στις 30 Μαΐου στη Μητρόβιτσα συνέβη αυτό το περιστατικό και χάρη στην δράση της αστυνομίας, της τοπικής αστυνομίας, ε, ξεκαθαρίστηκε το τοπίο. Όλοι αναγνωρίζουν ότι η αστυνομία του Κοσμοπεδίου κάνει καλή δουλειά. Ε, το βασικό λοιπόν είναι να σας και να στείλουμε περισσότερους δικαστές. Πέστε μας τι μπορούμε να κάνουμε. Κάτι που είναι προβληματικό και που ήταν ακόμη πιο προβληματικό πριν να αρχίσετε να διερευνάτε τις υποθέσεις διαφθοράς είναι η υπόθεση του Άλμπιν Κούρτε. Σκοτώθηκαν δύο άτομα και ο κύριος Κούρτε θα εμφανιστεί στο δικαστήριο για να καταθέσει. Ε, αρνείται την ε, νόμιμη παρουσία της Γιούλεξ, δεν θεωρεί ότι είναι τμήμα του τοπικού δικαστικού συστήματος. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ακόμη και όσοι δεν συμμερίζονται τις πολιτικές πεπιθήσεις του Κούρτε, τον υποστήριξαν σε αυτές τις αμφισβητήσεις που έχει απέναντι στη Γιούλεξ. Υπάρχει κάποιος τρόπος χάρη στον οποίο αυτή η στάση του Άλμπιν Κούρτε μπορεί να σταματήσει. Γιατί δεν βοηθάει την εικόνα της Γιούλεξ. Δύο Ρουμάνοι αξιωματικοί σκότωσαν αυτούς τους ανθρώπους, αλλά ακόμη είναι ελεύθεροι, δεν έχουν παραπευθεί στη δικαιοσύνη, ενώ ο κύριος Κούρτε ε, δικάζεται για κάτι το οποίο λέει ότι ήταν αρχικά μια διαδήλωση, όμως που εξελίχθηκε σε βίαιη διαδήλωση. Ε, η στάση και οι δηλώσεις του Κούρτε δεν βοηθούν την ε, εικόνα της Γιούλεξ. Εγώ αναγνωρίζω βέβαια την εξαρτησία του δικαστικού κλάδου, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το, την πολιτική διάσταση. Για τους Ρουμάνους ε, που συμμετέχουν στο προσωπικό της Γιούλεξ. Δύο αστυνομικοί Ρουμάνοι της Γιούλεξ ε, συνελήφθησαν να κάνουν λαθρεμπόριο τσιγάρων. Τι συμβαίνει με αυτούς. Είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τους δικάσουν για αυτή τους την πράξη. Γιατί αν εμείς ζητάμε να εφαρμόσει το κράτος δικαίου το κοσφοπέδιο, ενώ τα δικά μας κράτη-μέλη δεν κάνουν τίποτα, δεν έχει νόημα. Πρέπει και εμείς να είμαστε αξιόπιστοι και να είμαστε αυστηροί απέναντι στα εγκλήματα. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα μείζον έγκλημα, ένα παράπτωμα, γιατί κάνουν λαθρεμπόριο τσιγάρων, όχι όπλων. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πάνε στο δικαστήριο. Τι θα συμβεί με αυτό. Για το Βορρά τώρα, και εδώ σας συγχαίρω που προσπαθείτε να είσαστε πιο παράοντες. Ε, επισκέφθηκα το γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συναντήθηκα με τον ε, πρέσβη Τσιφώνη. Υπάρχει πρόοδος, αλλά μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα. Έγινε στη Μητροβίτσα μία διάσκεψη τέλος Μαΐου που την διοργάνωσαν οι Αλβανοί και Σέρβοι του Κοσμοπεδίου με θέμα διαιρεμένες πόλεις. Ε, προσπάθησαν να δουν τι μπορούν να κάνουν μαζί. Ο κόσμος ήρθε μέσω του Βελιγραδίου και της Πρίστινα. Ε, κάναν μια θαυμάσια δουλειά για να δείξουν ότι οι Αλβανοί και οι Σέρβοι του Κοσμοπεδίου θέλουν να συνεργαστούν. Παρότι δεν τους αρέσει ας πούμε, το, το πώς δημιουργήθηκε η κατάσταση, είναι διατεθειμένοι να δουλέψουν μαζί. Ακόμα μία ερώτηση. Τι γίνεται με το πρωτόκολλο των τελωνίων. Υπάρχει κάποια πρόοδος. Τι θα συμβεί σε αυτόν τον τομέα. Και κάτι τελευταίο πιο γενικό. Μετά από αυτά που είπε ο κύριος, λαμβάνω και αυτά που είπε ο κύριος Ντανζό. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας ε, από την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη εμφανίζεται με πάρα, πολλές, με πάρα πολλά πρόσωπα και φορείς και συχνά ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ποια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λένε ποιοι είναι αυτοί οι τύποι. Μήπως ε, με, την Ευρωπαϊκή, με την υπηρεσία αυτή εξωτερικής δράσης θα υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή ε, στις πολιτικές ε, και στην εικόνα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θα είναι ένας φορέας συγκεκριμένος, όχι πολλοί. Κάτι που είναι προβληματικό. Λόγω του προβληματικού καθεστώτος του κοσφεποδίου. Υπάρχουν τρία διαφορετικά νομικά συστήματα. Οι δικαστές που δουλεύουν με τη Γιούλεξ θα πρέπει να διαλέγουν ανάλογα με την ε, υπόθεση που εκδικάζουν. Τι επιπτώσεις υπάρχουν για τη δουλειά τους. Νομίζω ότι θα πρέπει ε, τα κράτη-μέλη να έχουν και αυτά πιο κοινή προσέγγιση. Και αυτό είναι σημαντικό. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορούμε ήδη να έχουμε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα και μετά υπάρχουν τέσσερις ομιλητέ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Χάουερ και στον κύριο Κέρμαμπον για να απαντήσουν τον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, θα κάνω μια πιο γενική προσέγγιση και ο κύριος Κερμαμπών θα σταθεί στα ιδιαίτερα ζητήματα τα οποία τέθηκαν σε σχέση με το ποιε είναι οι σχέση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, Όπως είπε και ο κύριος Κερμαμπών, επιτοπίως οι σχέσεις είναι οι καλύτερες δυνατές. Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο πραγματιστικής συνεργασίας, το οποίο είναι πολύ ψηλό, που καλύπτει και πάρα πολλά θέματα, όπως μπορεί να σας αναφέρει πιο λεπτομεριακά ο κύριος Κέρμαμπον, Υπάρχουν άλλοι χώροι βέβαια όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ πρέπει ακόμα να βελτιώσουν τη συνεργασία του Παραδείγματο χάρη στο Αφγανιστάν κάνουμε πολλές προσπάθειες για να βρούμε και εκεί χώρους δράσης που να είναι κοινοί. Χώρους δράσης που να είναι συμβατοί με τι εντολές και των μεν και των δε. Προσπαθούμε λοιπόν να ξεπεράσουμε τον απλό συντονισμό και την συμπληρωματικότητα και να περάσουμε σε χώρους κοινού συμφέροντος που να συνάπτονται και να είναι συμβατοί με την εντολή μας. Νομίζω ότι όλα αυτά εγγράφονται απόλυτα στο πνεύμα των επικεφαλής των φορέων μας να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτή την πραγματιστική συνεργασία Δεν θέλω τώρα να σταθώ βέβαια σε πολιτικά ζητήματα σε ό,τι αφορά την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εκπροσώπησή της λόγω της συνθήκης της Λισαβόνας προκύπτουν ορισμένες επιπτώσεις και η κυρία Άστιν έχει συζητήσει και με τους υπουργούς εξωτερικών για τα θέματα αυτά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης έχει συζητήσει με την κυρία Άστον δεν θέλω να στι λεπτομέρειε, θα αναφερθώ μόνο σε μία πτυχή η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική πάντα στα Βαλκάνια. Είναι οι διπλές αρμοδιότητες. Γιατί εκεί έχουμε μια κατάσταση κατά κάποιο τρόπο διπλού καπέλου, διπλών αρμοδιοτήτων, αρμοδιότητες εναντί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εναντί της διεθνούς κοινότητας. Και αν θέλετε θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπον. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματά σας, αλλά θα αναγκαστώ να λιγάκι συνοπτικός, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία έχετε ρωτήσει. Επανέρχομαι σε αυτά που είπε ο πρόεδρος στα εναρκτήρια σχόλιά του. Δεν θέλουμε να είμαστε θεαματικοί, θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και να ακολουθούμε μια πολιτική μικρών βημάτων. Αυτές είναι οι οδηγές αρχές της δράσης μας στο κοσφοπέδιο. Είμαστε εκεί όχι για να είμαστε στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, αλλά προωθήσουμε τη σταθερότητα στο κοσφοπέδιο για να βελτιώσουμε την κατάσταση εκεί και να αναλάβουμε τις ευθύνε μας. Έρχομαι τώρα στα διάφορα θέματα συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Φυσικά δεν μπορώ εγώ να αναφερθώ στα πολιτικά θέματα. Αυτό το οποίο είναι απαραίτητο, όπως ελέγχθη, είναι το να εξασφαλίσουμε κάτι το πρωταρχικό, να μπορέσουμε να βρούμε κοινού τρόπους δράσης για να διατηρήσουμε την ασφάλεια και τη σταθερότητα στο κοσυφοπαίδιο. Είμαστε προσιλωμένοι σε αυτή την κατεύθυνση από την αρχή και μπορώ να σας δώσω μερικά πρακτικά παραδείγματα. Έχουμε ξεκινήσει με την προσέγγιση για τρεις κοινέ δράσεις. Καταρχήν η αστυνομία του κοσυφοπαιδίου, γιατί αυτοί θα πρέπει να έχουν τις πρώτες δράσεις το τις Αν δεν τα καταφέρουν, εάν τους ξεπεράσουν τα πράγματα, τότε η ULEX σε συνεργασία με την εκτελεστική εξουσία με τις μονάδες διατήρησης της τάξης θα πρέπει να παρέμβει και αν τα πράγματα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα και χρειαστεί χρήση πυροβόλων όπλων, έρχεται η K4 να συμμετάσχει. Είναι δύσκολα όλα αυτά βέβαια να εφαρμοστούν γιατί χρειάζονται συνεδριάσεις συντονισμού, να υπάρχουν επαφές μέσω αξιωματικών συνδέσμων και κοινέ ασκήσεις ώστε να υπάρχει πλήρης συντονισμό ώστε να αποφύγουμε να μην ξαναγίνει αυτό που είχε γίνει το Μάρτιο του 2004 επειδή δεν υπήρχε αρκετό συντονισμός. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και νομίζω ότι με όλες αυτές τις διαδικασίες έχουμε πολύ καλά παραδείγματα για να τα χρησιμοποιήσουμε στις περιπτώσεις αυτές όπου πρέπει να συνδυάζονται πολιτικές δράσεις και στρατιωτικές ενέργειες για την εξασφάλιση της ασφάλειας. Κάτι ακόμα, νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό, να μην ανακατέψουμε πρόβατα με έγιες. Δεν μπορούμε να βάλουμε κάποιους να κάνουν κάτι που δεν μπορούν να κάνουν. Ένα στρατιωτικός δεν είναι αστυνομικός. Ένας αστυνομικός δεν είναι στρατιώτης θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία, θα πρέπει να υπάρχει συντονισμό, αλλά δεν θα πρέπει να ζητήσουμε από τη μία ή την άλλη συνιστόσα να κάνουν κάτι το οποίο είναι πέραν των ευθυνών και των δυνατοτήτων του. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνα. είμαι ο πρώτος ο οποίος θα τόνιζε την ανάγκη μιας απλοποίηση. Στο κοσκοπέδιο έχουμε πολλές ε, οργανώσεις που είναι παρούσες από, την, ε, από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο είναι απαραίτητο με αυτή την πλειάδα φορέων είναι να υπάρχει σαφήνεια για το ποιε είναι οι αρμοδιότητες του κάθε φορέα. Η ομάδα των Ηνωμένων Εθνών δίνει αυτή τη στιγμή την πολιτική κατεύθυνση στους ηγέτες των δυνάμεων καταστολής και επιβολής της τάξης, αλλά δεν δίνει λειτουργικές και επιχειρησιακές διαταγές, οι οποίες εξαρτώνται από τις ε, ε, επιτόπιες δυνάμεις. Αυτό είναι απαραίτητο για να υπάρχει λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα και η απαραίτητη υποστήριξη. Αυτό λοιπόν πρέπει να διατηρήσουμε και είναι ένα από τα σημαντικά στοιχεία είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορεί να είναι πάντα σαφής η κατανομή των αρμοδιοτήτων και μετά από την εφαρμογή της συνθήκης Λισαβόνας. Η Κομισιόν είναι ο τρίτος παίκτη. Είμαστε πάντα σε συντονισμό με την Κομισιόν γιατί πρέπει να εφαρμόσουμε σχέδια επιτοπίως τα οποία θα έχουν σαν στόχο να υποστηρίξουν τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διευκολύνουν τις δράσεις της ULEX. Για τα θέματα δικαιοσύνης. Υπάρχουν πολλέ προσδοκίες και έχουμε επίγνωση αυτού του γεγονότος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το Πασχοπέδιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχουν αυτές οι αποστολές. Αλλά θα πρέπει να έχουμε δύο βασικές αρχές στο μυαλό μας πάντα. Καταρχήν είναι πάρα πολύ ασθενικές οι δικαστικές αρχές στο Κωσικοπαίδιο. Ο αρχικός απολογισμός δεν ήταν καθόλου ικανοποιητικός. Με μία αποστολή υποστήριξης μπορούμε να τους βοηθήσουμε αλλά υπάρχουν και δράσεις που πρέπει να γίνουν από αυτούς τους ίδιους. Εμείς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τους νέους στο κοσμοπέδιο και να προετοιμάσουμε το μέλλον. Δεύτερον, η δικαιοσύνη είναι μια δικαιοσύνη η οποία καθυστερεί πάρα πολύ τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια, όπως και πολλές φορές στις χώρες μας. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα, οι δίκες που πρέπει να αντιμετωπιστούν και υπάρχει η πολιτισμική πτυχή, υπάρχουν άτομα τα οποία έρχονται από, πολιτικούς, από διαφορετικούς πολιτισμούς, πρέπει να ληφθεί απόψη το γεγονό ότι έχουν διαφορετικέ εμπειρίε, υπάρχουν πάντα τα προβλήματα του να βρουν του απαραίτητου μάρτυρες για να υπάρχουν τα αποδεικτικά στοιχεία για τη διεκπαιρέωση των, <clears throat> των δικογραφιών κτλ. Πρέπει λοιπόν να είμαστε λογικοί σε σχέση με το τι είναι εφικτό και ότι όχι. Νομίζω ότι όπως είπα και στην αρχή, είμαστε σε μια κατάσταση όπου έχουμε καλύτερο έλεγχο για όλα αυτά τα θέματα και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε χωρίς να παρέμβουμε στη λειτουργία των ανεξαρτήτων αρχών. Αυτό είναι μία από τις αρχές που θέλουμε εμείς να τονίσουμε, ότι πρέπει εμείς να μην παρεμβαίνουμε και να μην περιορίζουμε την αυτονομία της ε, εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής αρχής στο κοσμοπέδιο. Θα πρέπει εμείς απλώς να τους βοηθούμε να δώσουμε κι εμείς το καλό παράδειγμα και να μην δεχτούμε οποιαδήποτε παρέμβαση εκ των έξω. Κατά πόσο τώρα είναι σε κίνδυνο η σταθερότητα του κοσμοπεδίου, εγώ είμαι πεπισμένος ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο για τους λόγους που ανέφερα προηγουμένως. Υπάρχει μια μεγάλη προσδοκία για την δράση της Ιουλέξ, η οποία έχει συμβάλει τα μάλα στη σταθεροποίηση. Αλλά πιστεύω επίση ότι και η πολιτική του Κωσυφοπεδίου και ιδιαίτερα ο Πρωθυπουργό έχουν απόλυτη επίγνωση τη ανάγκη να υπάρξει σταθερότητα για να αντιμετωπιστεί και η διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα και γι' αυτό θέλουν να προχωρήσουν προ την κατεύθυνση αυτή με τον κάθε σεβασμό για τη σταθερότητα. Αυτό σημαίνει όμω ότι χρειάζεται την υποστήριξή μα. Χρειάζεται την υποστήριξη τη ULEX αλλά γενικότερα και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουν ότι τους υποστηρίζουν οι Βρυξέλλες, γιατί έχουν να περάσουν και δύσκολες στιγμές. Συνεχίζον στον τομέα αυτό, λέω πάντα ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Αυτό είναι μια σημαντική αρχή που πρέπει να την εφαρμόσουμε. Όσο εφαρμόζεται λοιπόν αυτή η αρχή, θα πρέπει να γίνει κατανοητή από όλους. σε ό,τι αφορά την έλλειψη προσωπικού, έχουμε πραγματικά σημαντικές ελλείψεις <clears throat> σε προσωπικό και συμφωνώ μαζί σας στο ότι η αστυνομία του Κωσυφοπεδίου είναι μια αστυνομία που λειτουργεί τώρα πολύ καλά παρά το γεγονός ότι ακόμα υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. Κάποια στιγμή θα μπορούσαμε να προβλέψουμε είναι κάπως πρόωρο να υπάρξει μια μεγαλύτερη ε, παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση των τοπικών δυνάμεων. Τόνισα ότι η προτεραιότητά μας είναι η δικαιοσύνη. Σας ανέφερα ποιε είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Έχουν ακόμα οξυνθεί λόγω της έλλειψης ε, εισαγγελέων και δικαστών. πολλές υποθέσεις οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Μα γι' αυτό εμείς ε, τονίζουμε πάντα στα κράτη-μέλη, έχετε εγκρίνει αυτή την ε, αποστολή με πάρα, πάρα πολύ φιλόδοξους στόχους, δώστε μας τα μέσα για να επιτύχουμε σε αυτή την ε, αποστολή και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα για την εσωτερική ασφάλεια στο κοσμοπέδιο, όλα αυτά που κάνουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε δίκτυα, λαθρεμπορίας ανθρώπων, πορνείας, λαθρεμπορίας όπλων, ναρκωτικών και όλα αυτά. Όλα αυτά για να μπορέσουμε να δράσουμε εναντίον τους είναι απαραίτητο να έχουμε τις απαραίτητες δικαστικές αρχές. Δεν θέλουμε εξάλλου να εξαχθούν και στις άλλες χώρες των Βαλκανίων. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε και μια πιο περιφερειακή αντιμετώπιση. Είναι απαραίτητο να μην εξαπλωθούν τα δίκτυα αυτά και προς την κατεύθυνση των δικών μας χωρών. Αυτό πρέπει να είναι ένα επιχείρημα που θα το κατανοήσουν τα κράτη-μέλη. Για τον Κούρτη, ναι, ναι, είναι σημαντικό αυτό που είπατε. Εγώ πιστεύω ότι και εκεί δεν πρέπει να υπάρξει παρέμβαση από τη δική μας πλευρά. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Θα πρέπει να παρουσιαστεί ενώπιον των δικαστηρίων για να επιληφθεί το θέμα αυτό, να ληφθεί υπόψη όλη η προβληματική από τα δικαστήρια. Όσο πιο γρήγορα επιληφθεί το θέμα αυτό, τόσο πιο ευτυχισμένοι θα είμαστε όλοι μας και τόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα. Για τους Ρουμάνους αλλά Αναφέρθηκε αυτό για τους δύο Ρουμάνους οι οποίοι συνελήφθησαν με λαθρέα προϊόντα, τσιγάρα αλλά και αλκοόλ. Εμείς είμαστε σε επαφή με τις Βρυξέλλες και τις Ρουμανικές Αρχές και δράσαμε αστραπία. Ε, απειλάγησαν από τα καθήκοντά τους αμέσως και απεστάλησαν στη Ρουμανία όπου υφίστανται αυτή τη στιγμή μια, μια έρευνα από τις εθνικές αρχές. Δεν μπορώ τώρα εγώ να προκαταλάβω τα συμπεράσματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί η ρουμανική αποστολή να κάνει μια εσωτερική έρευνα για να δει ποιοι είναι υπεύθυνοι για όλα αυτά τα οποία είναι και αναμένω ακόμα τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας στις επόμενες μέρες. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας με στεναρό τρόπο. Ξέρουμε ότι μια τέτοια, τέτοια ολιστήματα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην αποστολή μας και φυσικά δεν μπορούμε να τα αποδεχτούμε. Για το πρωτόκολλο σε σχέση με τα τελωνία. Προς το παρόν είμαστε σε στενή σε στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΟΗΕ Δεν είναι μονάχα θέμα λοιπόν της ULEX. Εμείς βασιζόμαστε σε ένα πλέγμα αρχών με στόχο να βρούμε τους τρόπους δράσης οι οποίοι θα μπορέσουν να εφαρμοστούν θετικά και αυτή τη στιγμή οι κοσοβαρικές αρχές μελετούν αυτό το πλαίσιο να δουν κατά πόσο μπορούν να δεχτούν αυτές τις αρχές και έχουμε επίσης ξεκινήσει κάποια διαβήματα έναντι του Βελιγραδίου για να δούμε αν και από εκεί μπορούν να γίνονται κτές αυτές οι αρχές. Ο στόχος είναι να υπάρξει πλήρης έλεγχο των τελωνίων σε όλο το κοσμοπέδιο και σε ό,τι αφορά το δίκαιο που εφαρμόζεται, που ήταν το τελευταίο σα ερώτημα, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο οφείλεται και στην κυριαρχικότητα και στο καθεστώ του κοσμοπεδίου. Αυτό είναι και αυτό αρμοδιότητα τη ULEX και ευθύνη τη. Εμείς έχουμε, μέχρι να διαλευκανθούν όλα αυτά, έχουμε δεχτεί ότι υπάρχουν τρία σημεία αναφορά στο το δίκαιο οι αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και το δίκαιο του Κοσμοπεδίου και οι δικαστές πάντα αποφασίζουν ποια από αυτές τις αναφορές ισχύει σε σχέση με την ημερομηνία διάπραξης ενός αδικήματος. Είναι μια προσωρινή λύση, φυσικά δεν είναι η οριστική λύση, αλλά αναμένοντα να υπάρξει μια οριστική λύση, αυτό είναι ο κανόνα τον οποίο εφαρμόσουμε. Σα ευχαριστώ, ήταν πλήρη η απαντήση σα. Και τώρα δεν μένει παρά δεν έχουμε παρά 12-13 λεπτά για τέσσερις ερωτήσεις. Παρακαλώ λοιπόν να είστε όλοι σύντομοι και όλες σύντομες. Η κυρία Κοπά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κλόμπενχάουερ, κύριε Ντεκερμαμπών. Νομίζω ότι η επιτυχία της Γιούλεξ είναι ακριβώς ότι την υποστηρίζουν όλα τα κράτη-μέλη και όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Και είναι πολύ σωστή αυτή η προοδευτική εφαρμογή που κάνει η Γιούλεξ αρχίζοντας από τη Μητρόβιτσα. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί ένα αίσθημα εμπιστοσύνης στους ε, τοπικούς παράγοντες. Η αστυνομική συνεργασία μεταξύ Γιούλεξ και Σερβίας ήταν επίσης ένα πρόσθετο θετικό βήμα. Θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήματα λοιπόν και στους δύο. Πρώτον, Ξέρουμε ότι τώρα έχουμε έναν σύνδεσμο στο Βελιγράδι. Αυτή η συνεργασία με τη Σερβική Αστυνομία τι ακριβώς σημαίνει στην πράξη και πώς την αξιολογείται μέχρι τώρα. Δεύτερον, για το Περιφερειακό Δικαστήριο της Μητροβίτσης. Ξέρουμε ότι η Γιούλεξ κάνει την προσπάθεια να το διοργανώσει, δεν αρκεί βέβαια μέχρι τώρα θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε ποια κατάσταση επικρατεί εκεί. Το προσωπικό του δικαστηρίου αυτού σε δικαστές και δικηγόρους και εισαγγελείς είναι αρκετό τέλος. Χάρηκα ιδιαίτερα όταν άκουσα αυτά που κάνετε για την προστασία ορισμένων Ορθοδόξων μοναστηριών που ενδιαφέρουν μερικές χώρες μέλη και μερικές χώρες της περιοχής. Ευχαριστούμε κύριε Στέλλερ. Δύο ερωτήματα ήθελα να θέσω. Πρώτον, για τη διαφθορά. Πρώτο το θέμα των ε, υποψιών για διαφθορά που αναφέρθηκαν σε σχέση με την κυβέρνηση του Θάτση. Αυτό ίσως θα ήταν και η Λιδία Λίθος σε σχέση με την πολιτική οριμότητα της κυβέρνησης ε, Θάτσι, Ποιες είναι οι συγκεκριμένες περιπτώσεις που χρειάστηκε να αντιμετωπίσετε και ποια είναι τα συγκεκριμένα βήματα στα οποία προβήκατε σε σχέση με τα θέματα της ε, διαφθοράς στον κυβερνητικό τομέα. Εμείς φυσικά υποστηρίζουμε πλήρως αυτήν την ε, αποστολή και ως Κοινοβούλιο μας ενδιαφέρει να ξέρουμε και σε ποιο βαθμό αυτές οι ενέργειες έχουν υποστηριχθεί δεόντως από τα κράτη-μέλη με την παροχή του αντιστοίχου προσωπικού. Ένα δεύτερο ερώτημα. Μιλάτε για, την, ε, για το διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων <clears throat> μεταξύ στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων. Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά μικτές ενέργειε και στρατιωτικού και στρατιωτικού χαρακτήρα. Και η, το ΝΑΤΟ έχει μια καλή εμπειρία για όλα αυτά τα θέματα, έχει χρησιμοποιήσει σώματα όπω η Ιταλοί καραμπινιέροι για να αντιμετωπίσει τέτοιου είδου αποστολέ. Ποια είναι τα συμπεράσματα τα οποία εσείς μπορείτε να αντλήσετε ε, ώστε να δώσετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα να λειτουργήσει σε πιο αποτελεσματικό τρόπο με τις ε, δυνάμεις αυτές Ξέρουμε λοιπόν ότι υπάρχει το παράδειγμα αυτό της Ιταλίας που έχει δυνάμεις οι οποίες μπορούν να παίξουν τους δύο αυτούς ρόλους, αλλά τι θα μπορούσατε να κάνετε στην Ευρώπη για να, στην Ulex να γίνεται με πιο ε, αποτελεσματικό τρόπο. Η Άννα Γκόμες. <clears throat> Χαίρομαι με την εξέλιξη που έχετε περιγράψει στο Κωσυφοπαίδιο και χαίρομαι γιατί αυτή η εξέλιξη την χάνει θετικής αναγνώρισης έτυχε μάλλον θετικής αναγνώρισης από τον Υπουργό Άμυνας της Σερβίας, εξωτερικών της Σερβίας, στην ομιλία του στο Συμβούλιο ασφαλεία. Είναι πολύ θετικά ότι υπάρχει αυτή η νέα προσέγγιση και από τη μεριά της Σερβίας που είναι χωρίς καμιά αμφιβολία αποτέλεσμα της προσέγγισης που ανέπτυξε η UNEX. Συμφωνώ ότι έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό σταθερότητα, αλλά το ερώτημα το επόμενο είναι η υποστήριξη που βρίσκεται για, το, για την εδραίωση του κράτους δικαίου. Είναι πολύ σημαντικό ότι η ULEX ξεκίνησε να είναι πολύ ενεργή στην αντιμετώπιση της <clears throat> διαφθοράς που είναι βασικό στοιχείο για την επίτευξη κράτους δικαίου. Αλλά υπάρχει μια άλλη πλευρά στο Κωσυφοπαίδιο η οποία έλειπε την τελευταία φορά που ήμουν εκεί το 2008 ήταν η οικονομική συνιστόσα. Το ερώτημα μου είναι τι κάνει η οικονομία για την ατμήμα της διαφθοράς οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό σε ό,τι αφορά αυτά που έκανε ή δεν έκανε η UNMIC σε ό,τι αφορά την ανάνυψη της οικονομίας ή την, απο... ή την αποτυχία ανάνυψης. Τι έγινε με το σταθμό παραγωγής ηλεκτρισμού, τι έγινε με άλλες πηγές εισοδήματος δυνητικά που θα μπορούσαν να υπάρχουν και να, ώστε να μην αναγκάζονται οι άνθρωποι να περνάνε στη μαύρη οικονομία, που είναι η πραγματικότητα τουλάχιστον το 2008 για το Και το άλλο μου ερώτημα είναι το εξή. Υπήρχε στο παρελθόν ένα πρόβλημα όχι μονάχα με την εθνοτική σερβική ε, μειοψηφία, αλλά και για τους Ρωμά σε ορισμένες περιοχές. Πώς αντιμετωπίζετε το θέμα αυτό. Και το θέμα των γυναικών, βέβαια. Δεν υπήρχαν αρκετές θέσεις ε, θέσεις ευθύνης. Κανένας από τους πρεσβευτές, παραδείγματος χάρη, δεν είναι γυναίκα. Και οι γυναίκες του Κοσφοπεδίου που οργανώθηκαν από τη UNICEF ήταν οι πρώτες οι οποίες φέρανε στη γνώση μας τα θέματα της ε, διαφθοράς. Και τόνισαν ότι ο λαός του Κοσφοπεδίου περιμένει να υπάρχει ένα αγώνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διαφθορά μα. Αν δεν το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιο θα το κάνει. Γιατί το ιστορικό τη UNMIC για αυτό το θέμα είναι πολύ αρνητικό. Τελευταίο ερώτημα. Ποια είναι η άποψή σα για το εξή. Ελέγχθη ότι υπάρχει μια αίτηση για αύξηση προσωπικού στο γραφείο της ανώτατης ε, εκπροσώπου στην, ε, στο Κωσυφοπέδιο και άνοιγμα ενός γραφείου στο Βελιγράδι. Γιατί θέλετε να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί έχουμε ήδη ένα γραφείο του ΟΗΕ εκεί. Ο κ. Κέλλομ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε την επιτυχία της Ulex. Α, μας ικανοποίησε το μήνυμα που μας στείλετε και η εμπειρία που έχετε αποκομίσει. Ε, αυτό που μας λέτε για την έλλειψη επαρκούς προσωπικού ε, στη Ulex. Πιστεύω ότι το άκουσαν οι ευρωβουλευτές και θα το διαβιβάσουμε στις κυβερνήσεις μας. Μία ερώτηση για το ρόλο της ε, κοινωνίας των πολιτών στο κοσφοπέδιο. Υπάρχει περίπτωση η Γιούλεξ να συνεργαστεί περισσότερο ή να υποστηριχθεί από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Κάτι που ανέφερε και η κυρία Αναγκόμες. Για πιθανές εντάσεις μεταξύ των ε, κοινοτήτων. Και ποιες είναι οι πηγές αυτών των εντάσεων. Μιλάω για Αλβανούς και Σέρους που μπορεί να έχουν διαφορές. Σίγουρα θα υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες από τις διάφορες κοινότητες των, της πρόσφατης ιστορίας και τις τραγωδίες που συνέβησαν. Και έπειτα, οι έρευνες στον Υπουργό Μεταφορών Οι απλοί Κωσοβάροι, τι άποψη έχουν για αυτές τις έρευνες. Οι υπόλοιπε υπηρεσίε, οι υπόλοιποι φορεί διδάχτηκαν κάτι, θεωρήθηκε επιτυχία αυτή η προσπάθεια. Ευχαριστώ. Και τώρα οι απαντήσεις. Um, yes, thank you, Chairman. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς όλους εσάς γιατί εκφράσατε την υποστήριξή σας των Αποστολών, ιδιαίτερα δε των εργασιών τους. Καθώς και σας ευχαριστώ για την δήλωση ότι θα μεταφέρετε στις κυβερνήσεις σας και τους εθνικούς σας συναδέλφους τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε για το προσωπικό. Αυτό ισχύει και για άλλες αποστολές βέβαια, αλλά θα μας βοηθούσε ιδιαίτερα. Η διαφθορά στη Γιούλεξ βέβαια το θέμα της διαφθοράς το αντιμετωπίζουμε από αστυνομική άποψη. Γίνονται προσπάθειες και από άλλους στην Κομισιόν και άλλα μέλη της διεθνούς κοινότητας για να μειωθεί η διαφθορά και οι δυνατότητες δωροδοκίας μέσω αδιαβλήτων διαδικασιών και του σεβασμού ορισμένων κανόνων. Οι δημόσιες προμήθειες είναι νομίζω ένα ιδιαίτερο ευαίσθητο θέμα εδώ. Η μικροδιαφθορά όμως, οι μικροδοροδοκίες ή τα μπαξίσια δεν σημειώνονται σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό στο κοσυφοπέδιο, έχουν μειωθεί ήδη. Ως προς αυτό το πρόβλημα λοιπόν, κυρίως η μεγαλοδιαφθορά είναι και η μεγαλοδοροδοκία. Βέβαια στην ουσία αυτό ξεπερνάει την εντολή μας, αλλά το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι κάθε φορά που πηγαίνω στην Πρίστινα βλέπω ότι είναι μία ανθυρή πόλη. Οι οικοδομικές δραστηριότητες αυξάνονται, δεν σημειώνονται φοβερές κλοπές, προχωράνε τα πράγματα, προχωράνε για το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών. Είχαμε κάνει μια μεγάλη συνάντηση τοπικών παραγόντων και μη κυβερνητικών οργανώσεων για να δούμε πώς ακριβώς θα οργανώνονταν τα πράγματα και ζήτησαν όλοι περισσότερη διαφάνεια και συνεργασία της κοινωνίας των πολιτών. Και αυτό προχωράει και αυτό. Και τέλος, τι γίνεται με τις έρευνες του Υπουργείου Μεταφορών. Μεγάλη λαϊκή υποστήριξη σημειώθηκε. Και όλοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τελικά εν καιρό το δέοντι και εν ευθέτω χρόνο θα διορθωθούν τα πράγματα. Να, αυτά. Ευχαριστώ. Σύνδεση. Η σύνδεση με το Βελιγράδι, ο σύνδεσμός μας με το Βελιγράδι είναι μόνιμος με την σερβική αστυνομία αλλά και με τα τελωνία και δικαστικούς κύκλους. Αυτό είναι απαραίτητο. Ναι και ο σύνδεσμός μας στο Βελιγράδι διευκολύνει την οργάνωση επαφών και μεταφορά, μετάδοση, υποβολή πληροφοριών κλπ. και από τις δύο πλευρές. Είναι πολύ καλή λοιπόν αυτή η συνεργασία, οι διαδικασίες που εφαρμόζονται είναι σωστές και σας επαναλαμβάνω αυτό που σας είπα και πριν. Είναι τεχνικό θέμα και πρόκειται για κοινό συμφέρον, τα ίδια συμφέροντα έχουμε με τη Σερβία κατά πολέμηση του οργανωμένου τους και της διαφθοράς. Καθώς και σε άλλους τομείς ας πούμε. Όταν οργανώνονται σημαντικά, οργανώνεται κάτι σημαντικό στο κοσυφοπέδιο όπως επίσημες επισκέψεις ένας από τους δύο διευθυντές της αστυνομίας του Κωσυφοπεδίου είναι Σέρβος και βρίσκεται σε μόνιμη σύνδεση με την σερβική αστυνομία, με την αστυνομία της Σερβίας και έτσι τέτοια συνεργασία έγινε και κατά το, την ενθρόνηση του νέου Πατριάρχη Και γι' αυτό θα θέλαμε να υπογραφούν και άλλες δύο συμφωνίες συνεργασίας. Για το δικαστήριο της Μητροβίτσης τώρα, εδώ αρχίσαμε από το μηδέν. Τα πράγματα έχουν προχωρήσει αλλά όχι αρκετά γιατί δεν υπάρχουν τοπικοί δικαστές. Πήγα στο Βελιγράδι πριν από τρεις μήνες και κατάφερα δύο Σέρβοι δικαστές που είχαν φύγει από εκεί να επανέλθουν Έπεισα και τον πρόεδρο του Κωσφοπεδίου, Έγιναν και υποβολές και άλλων προτάσεων ονομάτων. Πάντως τελικά θα υπάρξουν δύο Σέρβοι δικαστές στο δικαστήριο της Μητρόβιτσας. Αν θέλουμε όμως να γίνουν αποδεκτοί πρέπει να έχουμε τη συμφωνία του Βελιγραδίου. Αυτό το πετύχαμε σχετικά γρήγορα. Τώρα, την συνεργασία ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το αν υπάρχουν δυσκολίες σε στατιωτικό και πολιτικό επίπεδο. Ε, σε ό,τι αφορά τις στρατιωτικές και τις πολιτικές επιχειρήσεις, αυτό που είναι σημαντικό είναι να προχωρήσουμε σε κοινό σχεδιασμό και συντονισμό επιτόπου. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Και για τη συνθήκη της Λισαβόνας ελπίζω ότι θα μας επιτρέψει ε, να, υπάρχει, να υπάρξει καλύτερη συνεργασία των ε, επιχειρήσεων των στρατιωτικών με τις πολιτικές. Και αυτό που κάναμε στο Κοσφοπέδιο μπορεί να χρησιμεύσει ως αφετηρία για προβληματισμό. Ε, ας πούμε οι καραμπινιέροι, οι, οι στη Γαλλία, οι χωροφύλακες στη Γαλλία, ε, η στρατιωτική αστυνομία, ε, τέτοιες ε, δυνάμεις θα μας ε, βοηθήσει να βρούμε μια σωστή ισορροπία μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών επιχειρήσεων, οικονομία και εκπαίδευση. Έχω απαντήσει ουσιαστικά η δημιουργία ενός κράτους δικαίου συνδέεται με την οικονομική πρόοδο και τις επενδύσεις. Είναι ένας κύκλος. Ε, όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Σε ό,τι αφορά τις εθνικότητες, ε, σερβικές, βοσνιακές, Ρώμα και Το θέμα δεν είναι για μας Δηλαδή η αποστολή μας δεν είναι να βελτιώσει τη μοίρα τους, αλλά να υπάρξει ασφάλεια συνολικά. Αυτό που μπορώ να πω για τις ε, μειονότητες είναι ότι δεν υπάρχουν εντάσεις μεταξύ των κοινοτήτων. Δεν υπάρχουν ε, πραγματικές απειλές ε, για την ελευθερία κίνηση. Υπάρχουν βέβαια ψυχολογικά εμπόδια δεδομένου του παρελθόντος. Υπάρχει πρόβλημα, ας πούμε, πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας το χώρο οι, τα μέλη των διαφόρων ε, ε, μειονοτήτων και οι Ορθόδοξοι κυκλοφορούν ελεύθερα στο κοσφοπέδιο. Σε ό,τι αφορά τη μοίρα των γυναικών, έχουμε ένα τμήμα για το φύλλο και τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, στο εσωτερικό της Γιούλεξ που είναι σε επαφή στενή όχι μόνο με τις διάφορες μη κυβερνητικέ οργανώσεις αλλά και πιο συγκεκριμένα με μη κυβερνητικέ οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα γυναικών και στην εντολή μας αναφέρεται συγκεκριμένα η εξασφάλιση του, της, των δικαιωμάτων και της ασφάλειας των πολιτών. Γι' αυτό ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών είναι πολύ σημαντικό και θέλουμε να έχουμε μονίμως ε, στενές σχέσεις με τις οργανώσεις της. Και μάλιστα εκδόθηκαν πρόσφατα κάποιες εκθέσεις από μη κυβερνητικές οργανώσεις που ήταν πολύ α, θετικές για τη στάση της Γιούλεξ. Και ο πληθυσμό μας υποστηρίζει. Όπως ε, υπόθηκε υπάρχει μεγάλη προσδοκία για το τι μπορούμε να πετύχουμε εκεί στο κοσμοπέδιο. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα της α, διαφθοράς και της καταπολέμησης της ε, διαφθοράς και του ρόλου μπορεί να παίξει η Ιούλεξ. Σας ευχαριστώ Ταμάλα για την παρουσία. Ένα στοιχείο το οποίο το λέω παρενθετικά. Μιλήσαμε πολύ για δικαιοσύνη, μιλήσαμε πολύ για διαφθορά. Αναφερθήκατε στους αγνοούμενους επίσης και για τα εγκλήματα πολέμου, τους αγνοούμενους κτλ. Και το ψυχολογικό κλίμα το οποίο επικρατεί και το οποίο πολλές φορές είναι πολύ διαφορετικό από τις προκαταλήψεις που ισχύουν για αυτούς που ατενίζουν το κοσμοπέδιο από τα έξω. Υπάρχουν δηλαδή συνδέσεις μεταξύ εθνοτικών ομάδων και δεν είναι τόσο στεγανά τα πράγματα όπως τα παρουσιάζουν μερικές φορές για την Πρίστινα και το Βελιγράδι, αλλά το θέμα των αγρογμένων είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε ένα είδος εμπιστοσύνη και επίση και την αξιοπρέπεια στην κοινωνία του Πεδίου, που είναι μια τραυματισμένη κοινωνία μετά από τα πρόσφατα γεγονότα. Αυτά που έγιναν λοιπόν με τη συνεργασία της Γιούλεξ και των αρχών του Βελιγραδίου είναι πάρα πολύ θετικά. Νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε αυτή τη συνεργασία. Δεν είναι πάντα τόσο δύσκολα να βρούμε πού είναι η τάφη των αγνοωμένων και να εντοπίσουμε τα άτομα αυτά που έπεσαν θύματα. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την συμφιλίωση μεταξύ των εθνοτικών ομάδων. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό κουράγιο. Και θα περάσουμε τώρα στη Βοσνία. Παρακαλώ.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 Συνεχίζουμε τις εργασίες μας με την Βοσνία Ερζεγοβίνη. Θέλω να καλωσορίσω τον στρατηγό Τζον Μακκόλ, ο οποίος είναι ο διοικητής της επιχείρησης ε, είναι ο διοικητής της Αλφέας. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται ενώπιόν μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για την παρουσία σας λοιπόν. και έχουμε και τον στρατηγό Φέλλερ, ο οποίος είναι επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης της ULEX ε, στην, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Βοσνία. Ο στρατηγός Μακόλ θα παρουσιάσει την Αλθέα και μετά και ο Χάουερ και ο στρατηγός Φέλερ θα παρουσιάσουν τα αστυνομικά θέματα. Θα έχουμε λοιπόν όλες αυτές τις ενημερώσεις για να μπορέσουμε στη συνέχεια να ομαδοποιήσουμε και τις ερωτήσεις σας. Σας παρακαλώ στις ερωτήσεις σας να είσαστε συνοπτικοί ώστε να έχουμε μια πλήρη ανταλλαγή απόψεων μέσα στο χρονικό όριο το οποίο μας περιορίζει. Στρατηγέ μου, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα για να ανταλλάξω απόψεις μαζί σας για τα επιχειρησιακά θέματα της Αλθέας με την, με την άδειά σας Θέλω να κάνω κάποιες επιχειρησιακού χαρακτήρα παρατηρήσεις. Όπως ξέρετε εγώ διοικώ την Αλθέα γιατί είναι μια επιχείρηση Βερολίνου ΣΥΝ και εγώ είμαι υπεύθυνο για τις δραστηριότητες του ΝΑΤΟ στον τομέα αυτό μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η ΧΕΙΦΟΡ και τη στρατηγική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαι ο συντονιστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ΝΑΤΟ, είμαι ο συντονιστής του ΝΑΤΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα για τη Βοσνία Ζεγοβίνη που είναι αυτό που σας ενδιαφέρει. Ξέρετε πόσο δύσκολη είναι η πολιτική κατάσταση εκεί, πόσο μεγάλες είναι οι προκλήσεις. Εγώ δεν θα καλύψω αυτό το θέμα, όχι μονάχα γιατί αυτό είναι έξω των, από τους αρμοδιότητές μου. Θέλω να εστιάσω περισσότερο στην Αλθέα. Θέλω να πω ότι παρά τη δύσκολη πολιτική κατάσταση, η κατάσταση ασφαλείας οποίο παραμένει γαλήνια και σταθερή. Έχουμε ένα σταθερό περιβάλλον που έχει διατηρηθεί για πολύ καιρό οι τοπικοί φορεί επιβολή του νόμου και τη τάξη καταδεικνύουν την ικανότητά του να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Η Αλθέα είναι η πιο μακρά επιχείρηση στο χώρο αυτό. Ε, το 2004 ξεκίνησε με περίπου 5.000 προσωπικού, το 2007 ε, μεταρρυθμίστηκε και έχει μειωθεί ο αριθμός του προσωπικού σε περίπου 2.000 άτομα 7.000 συνολικά έχουν υπηρετήσει σε αυτή την επιχείρηση από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το συνολικό κόστος είναι περίπου 23 εκατομμύρια ευρώ. Οι κύριοι στόχοι μας είναι να παρακολουθήσουμε τη συνεχιζόμενη συμμόρφωση με τις στρατιωτικές πτυχές της Συμφωνία του Dayton, να συμβάλλουμε στην σταθερότητα, επί το οποίο να δώσουμε εκπαίδευση, κατάρτιση και δημιουργία ικανοτήτων στις στρατιωτικές δυνάμεις επί το οποίο, αυτό είναι κάτι στο οποίο θα σταθώ λιγότερο αργότερα, να συλλέξουμε πληροφορίες και να αντιμετωπίσουμε και κάποια υπολοιπόμενα καθήκοντα της συμφωνίας του, του Dayton. Επίσης, εμείς υποστηρίζουμε τις ε, δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην και δίνουμε και, εάν χρειαστεί, τη δυνατότητα εκένωσης περιοχών από υπηκός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία της ε, Αλθέας. Είναι μια επιχείρηση η οποία βασίζεται στη συλλογή πληροφοριών. Παίζει σημαντικό ρόλο το να έχει πλοκάμια τα οποία δίνουν πληροφορίες και έχουμε μια μεγάλη εμπειρία για τη συλλογή πληροφοριών. Ο συντονισμός λοιπόν γίνεται από πέντε κέντρα συντονισμού. Υπάρχει επίσης ένα αέρια παρακολούθηση από ειδικέ ομάδες και ομάδες που ασχολούνται με τα θέματα ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Το κέντρο μας είναι έξω από το Σεράγεβο. Έχουμε ένα πολυεθνικό τμήμα και επίσης μια αστυνομική δύναμη. Έχουμε και έφεδρους σε επιχειρησιακό επίπεδο. Έχουμε, έχουμε εφεδρίες πέραν του ορίζοντος τις οποίες διαμοιραζόμαστε με την K4 και υπάρχουν ε, συμφωνίες που μας επιτρέπουν να μετακινούμε κόσμο μεταξύ των δύο θεάτρων ε, παρουσίας. Υπάρχει επίσης συνειδητοποίηση των κοινών αυτών καθηκόντων που περιλαμβάνουν θέματα όπως ο έλεγχος και η αποθήκευση πυρομαχικών και όπλων, ο έλεγχος του εναέριου χώρου και του ηλεκτρομαγνητικού ε, φάσματος. Τέτοιοι στόχοι, τέτοια καθήκοντα τώρα έχουν ε, δοθεί στο Υπουργείο Άμυνας ενώ προηγουμένω ήταν το Υπουργείο Ασφάλεια. Και εμεί συνεχίζουμε λοιπόν αυτέ τι δραστηριότητε και δίνουμε πληροφορίε και συμβουλέ, Ο στόχο είναι να είναι αυτόνομη κάποια στιγμή η δράση των τοπικών Υπουργείων και να είναι εναρμονισμένα με τα παγκόσμια πρότυπα εστιάζουμε στην εκπαίδευση και στη δημιουργία ε, ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων της Βοσνίας αλλά και της Ερζεγοβίνης. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να υπάρξουν σταδιακά περισσότερες αναλήψεις καθηκάντων. Ο στόχος μας είναι λοιπόν να εξασφαλίσουμε και αυτά τα οποία είναι απαραίτητα σε επίπεδο κατάρτισης και της δυνάμεις της Βοσνίας Ερζεγοβίνης με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και του ΝΑΤΟ. Όπως με τις περισσότερες στρατιωτικές επιχειρήσεις, ένα από τα βασικά προβλήματά μας είναι να έχουμε αρκετά στρατιωτικές δυνάμεις. Πολλοί από αυτούς οι οποίοι συνεισφέρουν στα θέματα είπαν ότι θα μειώσουν σημαντικά τις δυνάμεις τους. Αυτό θα σημαίνει ότι θα, μειώσουμε, θα μειωθεί η δύναμή μας κάτω από τα ελάχιστα απαραίτητα. Γι' αυτό εμείς έχουμε προσεγγίσει άλλα κράτη και έχουμε ζητήσει να αναθεωρήσουν την θέση τους. Χαίρομαι που υπήρξαν θετικές ανταποκρίσεις από ορισμένους και έτσι θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε μέχρι τον Νοέμβριο του 2010 πλήρη επιχειρησιακή δύναμη. Τι θα γίνει επέκεινα του 2010, θέλω να πω τα εξής πρώτα στις 25 Ιανουαρίου το Συμβούλιο δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη, εάν αυτό είναι απαραίτητο, να υποστηρίξει τις προσπάθειες Βοσνίας Ζεχοβίτης να έχει τις απαραίτητες δυνάμεις ασφαλείας πέραν του 2010 και βάσει αυτών που προβλέπονται για τις δυνάμεις αυτές φαίνεται ότι θα υπάρξει μια μεγάλη μείωση εάν δεν υπάρξουν κατάλληλε δυνάμεις ως το τέλος του έτους. Η ελπίδα μου είναι και θα θέλαμε να έχουμε μια πολιτική κατεύθυνση για τα θέματα αυτά μέχρι το καλοκαίρι. Αυτά ήθελα να σας πω και είμαι έτοιμος να απαντήσω στα ερωτήματά σας. Ευχαριστώ κύριος Κλάμπενχάουερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί βουλευτές, θα σας πω δύο λόγια για την αστομική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία Ζεγοβίνη που ακούσατε ήδη κάποια πράγματα. Είναι η παλαιότερη αποστολή ΕΠΑ. Ξεκίνησε πριν από 7 χρόνια, 1η Ιανουαρίου 2003, με την εντολή να εγκαθιδρύσει μια αποτελεσματική αστυνομική δύναμη με βάση τις καλύτερες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές. Το, η εντολή μας έχει ανανεωθεί πρόσφατα και τρέχει μέχρι τον Ιανουάριο 2012 Εστιάζουμε τώρα στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς. Η δύναμη... Έχουμε αριθμού με 120 ανθρώπους από, τα... από 24 κράτη-μέλη, καθώς και την ε, Ελβετία, Ουκρανία και Τουρκία. Έχουμε τέσσερα περιφερειακά γραφεία με πραγματογνωμοσύνη αστυνομική και εισαγγελική. Επίσης έχουμε αναλυτικό δυναμικό, μπορούμε να κάνουμε αναλύσεις και έχουμε και μια προσωρινή αποθήκη, ένα προσωρινό γραφείο. Η πολιτική κατάσταση, παρότι είναι ευαίσθητη στην ε, Βοσνία Ερσεγοβίνη. εμείς ε, συνεχίζουμε το έργο μας και έχουμε πετύχει συγκεκριμένα επιχειρησιακά αποτελέσματα. Θα ήθελα να σας τονίσω ότι έγιναν δύο επιχειρήσεις τοπικά που είναι γνωστές μέσω του τύπου. Θέλω να τονίσω την υποστήριξη που δόθηκε σε δύο βασικές επιχειρήσεις επιβολής του νόμου ε, σε όλη την Βοσνία Ρεσεγοβίνη. Η επιχείρηση ΑΦΟΣ και η επιχείρηση Δίκτυο. Ο επόμενος ομιλητής θα σας αναφέρει περισσότερα. Έχουμε δημιουργήσει και ένα συντονιστικό φορέα της ε, αστυνομίας με σκοπό να συντονίζονται οι διάφορες αστυνομικές δυνάμεις στον χώρο της Βοσνίας Ερζεγοβίνη. Και χάρη στην επιχειρησιακή σχεδόν θα έλεγα παρέμβασή μας βοηθούμε να διαλύσουμε ε, τοπικά και διεθνή δίκτυα εγκληματικά τα οποία φτάνουν μέχρι και τις ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι η αποστολή μας έμεσα ε, συνεισφέρει στην ε, εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια συμφωνία συνεργασίας με τη Europol, ούτως ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε αυτόν τον τομέα. Ένα βασικό στοιχείο της επιτυχίας μας είναι η καλή συνεργασία και συντονισμός με τη διεθνή κοινότητα και κυρίως με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το επίπεδο θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τον στρατηγό Μακόλ με, για την καλή συνεργασία με την επιχείρηση Αλθέα. Η αποστολή μας έχει σαν να προετοιμάσει και με μια στρατηγική εξόδου γιατί η εντολή μας ε, δεν θα ξανανεωθεί μετά το 2011. Αυτή η στρατηγική θα λάβει υπόψη διάφορα στοιχεία. Καταρχά, τη συνολική παρουσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Βοσνία Ερζεγοβίνη και την πρόοδο που έχει σημειώσει η αποστολή μα. Επίση, σημαντικό είναι η στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα ενδυναμωθεί ε, και μέσα στο πνεύμα τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή αναπτύσσει ένα πρόγραμμα σε στενή συνεργασία με στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, ώστε να υπάρξει μια συνέχεια σε ορισμένα καθήκοντα, εάν η δική μας αποστολή, όπως αποφασίσει το Συμβούλιο, σταματήσει. Θα ήθελα τέλος να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τον ταξίαρχο Φέλερ για τη, την συνεισφορά της δικής του αποστολής στην ε, εφαρμογή του κράτους δικαίου στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημερίζω τα αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα οποία ευχαριστώ. Και εγώ θα είμαι διαθέσιμος για ερωταπαντήσεις ως προς τις αστυνομικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις διοργάνωσης της αστυνομίας για την καλύτερη τήρηση της ενόμου τάξεως στη Βοσνία αλλά και στην Ερζεγοβίνη η εντολή που μας δόθηκε και οι επιτεύξεις της αποστολής για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου κλίματος θα είναι το θέμα μου. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Όπως πάντοτε σε τέτοιου είδους παρουσιάσεις, τονίζω πάντοτε ότι συμμεριζόμαστε απόλυτα τους στόχους παρά το ότι μέχρι τώρα δεν είχε σημειώθηκε καμία τρομερή επιτυχία. Τα πολιτικά και άλλα εγκλήματα, οι δεχθεί ιδίω δεν έχουν πάντως αυξηθεί ιδιαίτερα. Θα ήθελα να σας περιγράψω γενικότερα την εντολή της αποστολής. Ήταν η πρώτη αυτή τέτοιου είδους αποστολή της Ένωσης και άρχισε πριν από 8 χρόνια. Χρειάστηκε προσαρμογές πολλές φορές λόγω των αλλαγών στη Βοσνία Ερζεγοβίνη αλλά και της ταύτισης νέων στόχων. Η αποστολή αυτή ακολουθεί την αποστολή του ΟΗΕ για την πρώτη οργάνωση αστυνομία στη Βοσνία και την οικοδόμηση θεσμικών οργάνων. Από το 2006 μειώσαμε το προσωπικό από 450 διεθνείς αστυνομικούς σε 200 και ταυτίστηκαν τρεις πρόσθετοι στόχοι για την σταθερότητα της περιοχής και την σταδιακή απομάκρυνσή μας. Την ε, μεταρρύθμιση της αστυνομίας, την καταπολέμηση του οργανωμένου και άλλων εγκλημάτων και την ενδυνάμωση της εσωτερικής και εξωτερικής λογοδοσίας της αστυνομίας. Για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος θελήσαμε να συνεννοηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και να συνεργαστούν στενότερα. Όπως γνωρίζετε υπάρχουν πολλοί τοπικοί παράγοντες που ενδιαφέρονται από την οργάνωση της ε, νόμου τάξεως στη Βοσνία. Το 8 εγκρίθηκαν δύο νομοσχέδια αστυνομικής μεταρρύθμισης και εκεί έληξε η εντολή αυτή. Τον Ιανουάριο φέτος αποφασίστηκε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας ιδιαίτερα στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Παρακολουθούμε, επιτηρούμε και συμβουλεύουμε τους εταίρους μας και με τον νέο αυτό στόχο μειώσαμε σε 130 το διεθνές προσωπικό ενώ ταυτόχρονα συνεχίζουμε να συλλέγουμε πληροφορίες. Το προσωπικό αποτελείται από αστυνομικού, τελωνιακούς, ειδικού για την μετανάστευση, λογιστές και αναλυτές καθώς και πολιτικούς συμβούλους και ειδικού για θέματα δημοσίων πληροφοριών. 250 τοπικός απασχολούνται εκεί. Όλοι είναι αποφασισμένοι να σεβαστούν την ευρωπαϊκή, τα ευρωπαϊκά πρότυπα που θέλουν να εφαρμόσουν στη χώρα τους. Τρεις χώρες παρετήθηκαν από την προσπάθεια ενώ οι 27 ενωσιακές και άλλες 6 συμμετέ συνέχισαν μέχρι το 2009. Σήμερα μόνο 20 χώρες μέλη της Ένωσης έχουν στείλει προσωπικό καθώς και η Ελβετία, η Τουρκία και η Ουκρανία. Τώρα για τη συμμετοχή των γυναικών περίπου 15% του διεθνού μας προσωπικού είναι θηλυκό και θα θέλαμε οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποτελέσουν υπόδειγμα. Μειώσαμε την παρουσία μας επιτοπίως μόνο στην Πάνια Λούκα, τη Μόσταρ και το Σεράγεβο, το Μοστάρ και το Σεράγεβο και θελήσαμε να καλύψουμε παρόλα αυτά το σύνολο της επικράτειας και της Ρεπούμπλικα Σέρψκα. Ιδιαίτερα σε επίπεδο εισαγγελιών και αστυνομίας. Έρχομαι στα επιτεύγματα. Συνεργαζόμαστε επιτυχώς τεχνικά με τους εταίρους μας για την καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος. Σημειώθηκε πρόοδος και στην αστυνομία και στον τομέα της ποινική δίωξης. Συνελήφθησαν σε σημασμένη κακοποιή και μεταρρυθμίστηκε ο ποινικό κώδικας. Καταπολεμούνται από διάφορες οργανώσεις η λαθρεμπορία, καταπολεμάται η λαθρεμπορία ναρκωτικών, ιδιαίτερα στην Ανατολική Βοσνία και η αστυνομία είναι διατεθειμένη να αντιμετωπίσει και ικανή να αντιμετωπίσει τις οργανωμένες μορφές του εγκλήματος κατεσχέθηκαν εκατοντάδες κιλών ηρωίνης, σκάνκ, που είναι μια ειδική μορφή μαριχουάνας, και κατεστράφει ένα εργαστήριο. Όλα αυτά με τις δικές μας συμβουλές και επιτήρηση. Δύο χιλιόγραμμα κοκαίνης έχουν επίσης κατασχεθεί μόλις πριν από δύο εβδομάδες και πάνω από 150 ύποπτοι συνελήφθησαν. Όλα αυτά βασίστηκαν σε συνεργασία μεταξύ όλων των περιφερειακών αρχών και των γειτονικών χωρών Σερβίας, Κροατίας και Μαυροβουνίου. Η καταπολέμηση της, του πλησίματος βρωμίκου χρήματος επίσης έχει σημειώσει προόδους. Οι τελευταίοι αριθμοί το επιβεβαιώνουν. Η καμπάνια για την καταπολέμηση της ε, αυθοράς έχει επίσης σημειώσει πρόοδο λόγω της λήψης νέων μέτρων. Τώρα η θεσμική ανάπτυξη έχει και αυτή προχωρήσει, αν και μερικές φορές πολύ αργά. οι ποινικέ διώξει δεν διχάνουν πάντα συμφωνίας μεταξύ των δύο οντοτήτων της Βοσινίας. Ο διάλογος, η συνεννόηση για τις θεωρήσεις προχωρεί. Τα Υπουργεία και η αστυνομία καθώς και οι πολίτες περιμένουν τις τελευταίες προτάσεις της Κομισιόν για την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Και τώρα οι μελλοντικές προκλήσεις, τελειώνω, τελειώνω τώρα, ρόλος μας θα συνεχίσει να είναι η σταθεροποίηση της κατάστασης και άρα η συμβολή στην σταθερότητα της περιοχής και ο συντονισμός με τη συνεργασία για την επιβολή της ενόμου τάξεως. Θέλουμε να υπάρξουν βιώσιμοι και σταθεροί μηχανισμοί για την καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος. Ταυτόχρονα θέλουμε να έχουμε απτά αποτελέσματα και παραλλήλως συνεργαζόμαστε στενά με την Κομισιόν και με τοπικές αρχές για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την προενταξιακή διαδικασία κυρίως μέσω της μεταφοράς πληροφοριών και γνώσεως ώστε προοδευτικά να, μπορέσουμε, να μπορέσουν όλοι οι, παράγον, οι ενωσιακοί παράγοντες να εναρμονίσουν τις προσπάθειές τους και να μπορέσει να καταλήξει η επιχείρηση επιτυχώς μέσω της εμβάθυνσης και ενδυνάμωσης της πολυπλευρής συνεργασίας. Να κάνω τρεις ερωτήσεις προς τον ε, στρατηγό Μακόλ πριν δώσω το λόγο στους αδέλφους. Πρώτον, ένα σχόλιο μάλλον, όχι ερώτηση. Για τις συνεχείς αξιολογήσεις του Συμβουλίου ή και άλλων που μιλούν για ένα περιβάλλον ε, ασφάλειας ως προς περιβάλλον ασφάλειας στη Βοσνία που δικαιολογούν την απόσυρση της ε, στρατιωτικής αποστολής. Συχνά έχουμε διαφορετικές ερμηνείες, αλλά πραγματικά διερωτώ αν έχει νόημα να διατηρήσουμε μια στρατιωτική δύναμη στη Βοσνία τώρα. Όταν ξέρουμε ότι ουσιαστικά οι δυσκολίες δεν έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, είναι περισσότερο πολιτικές και θεσμικές. Παρ' όλα αυτά επιλέγει η διατήρηση της αποστολής και η σταδιακή μετατροπή, ο σταδιακός μετασχηματισμός σε Εδώ έχουμε 2.000 άτομα εκεί. Α, πώς θα κάνουμε το μετασχηματισμό Πώς θα γίνουν αυτές δυνάμεις οι οποίες ασχολούνται με την κατάρτιση στρατιωτικού προσωπικού. Δεύτερον, η, οδός, η πρόοδος που κάνει η Βοσνία Ερσεγοβίνη προς το ΝΑΤΟ. Η πορεία της Βοσνίας Ερσεγοβίνης προς το ΝΑΤΟ. Πώς η επιχείρηση της Αλθέας μπορεί να ενσωματωθεί σε αυτή την προσπάθεια της Βοσνίας Ερσεγοβίνης να οδεύσει προς το ΝΑΤΟ. Τρίτον, Είπατε ότι η Αλθέα υποστηρίζει το δικαστήριο της Χάγης. Ο Χάτζιτς και ο Μλάδιτς δεν διώκονται ακόμα, δεν έχουν παραπευθεί στην, στην δικαιοσύνη. Κατηγορούνται για εγκλήματα που έχουν διεξάγει στην Βοσνία Ριζεγοβίνη. Πώς διεξάγεται η συνεργασία με το δικαστήριο. Τι εντολή έχει λάβει ως προς αυτό η επιχείρησή σας. Η κυρία Μπόσκουρτ. Ευχαριστώ. Θέλω να κάνω ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Καταρχάς, και εγώ πιστεύω ότι η αποστολή είναι πολύ σημαντική για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής. Είχα πάει στην περιοχή πριν από ένα μήνα και συνομίλησα με τους στρατιωτικούς. Ε, υπάρχουν άτομα που κατέχουν παράνομα όπλα εκεί. Όπλα τα οποία προέρχονται από το παρελθόν της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Έχεις Υπάρχει λοιπόν μια στρατηγική να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Τι θα κάνει η K4 για αυτό το θέμα, η U4 για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ κύριε Μπίτι Κόφερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ το στρατηγό ενημέρωση. Κύριε στρατηγέ μάλλον Μακόλ, διάβασα στο βιογραφικό σας ότι ασχολείται με ένα σπορ το οποίο θα μου άρεσε και εμένα. Τρέχω, αλλά με αργό ρυθμό. Πόσο αργό δηλαδή. Πολύ αργό. Πόσο αργός μπορεί να είναι κανείς. Όσο πιο αργός γίνεται. Ας σοβαρευτώ όμως τώρα. Στρατηγέ μου. για τη δύσκολη πολιτική κατάσταση. η οποία δεν έχει εκτραχυνθεί ακόμα. Δεν έχει επηρεάσει την ασφάλεια. Ευτυχώς. Από την εμπειρία που έχω, κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί όμως. Όταν μια κατάσταση είναι δύσκολη σε πολιτικό επίπεδο, συχνά υπάρχουν επιπτώσεις αρνητικές στον τομέα της ασφάλειας. Να θέσω λοιπόν το ίδιο ερώτημα που έθεσε και ο πρόεδρος, αλλά από διαφορετική σκοπιά. Μπορούμε να επιτρέψουμε στην Αλθέα να αποσυρθεί. Και σε περίπτωση που υπάρξουν προβλήματα ασφάλειας, ποιος θα είναι παρόν για να εξασφαλίσει την ε, ασφάλεια. Ποιος θα την αντικαταστήσει, αν θέλετε, την Αλθέα. Διακατέχουμε από μια κάποια απεσιοδοξία για την ε, μεμονωμένη απόφαση ορισμένων κρατών μελών να μην υποστηρίξουν πλέον την Αλθέα. Οι τελευταίες είναι η Ισπανία και η Ιταλία, που θα σταματήσουν τις δραστηριότητε τους. Είμαι αδαής βεβαίως. Και οι ερωτήσει μου ίσως είναι... Όχι ερωτήσει ενός επαΐοντα. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η Αλθέα θα εξασφαλίσει την ασφάλεια. Εσείς είπατε ότι ελπίζετε να το κάνει και όχι ότι περιμένετε να το κάνει. Και είπατε ότι Ελπίζετε ότι μετά το τέλος του 2010 θα συνεχίσετε την αποστολή σας. Τι χρειάζεστε για να περάσετε από την ελπίδα στην προσδοκία. Ότι δηλαδή η Αλθέα θα μπορέσει να τα καταφέρει και να εξασφαλίσει την ασφάλεια, παρότι αυτές οι δύο χώρες, Ισπανία και Ιταλία, αποφάσισαν να αποσυρθούν από την Αλθέα. Αυτή είναι η βασική μου ερώτηση. Έχουμε ευθύνη απέναντι στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Και γι' αυτό δεν πιστεύω ότι πρέπει να επιλέγουμε τη διαιώνιση κάποιων θεών περιοχών. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο ασφάλειας. και να υπάρχει και η απαραίτητη υποστήριξη. Δεύτερη ερώτηση, προς όποιον είναι αρμόδιος από τους ομιλητές. Για την ε, παρουσία δυνάμεων ασφαλείας από την Τουρκία στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Ένας συνάδελφος που πρόσφατα επισκέφθηκε τη χώρα μου είπε ότι η κυβέρνηση ανησυχούσε για το αν η Ευρώπη θα σεβαστεί τις εγγύησεις περί ασφάλειας. Τη στιγμή που η Τουρκία είπε ότι ό,τι και να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκείνη θα παραμείνει. Εσάς πώς, το, πώς σας φαίνεται αυτό. Είναι εταίρος σας, είναι ανεξάρτητη. Η Τουρκία βοηθάνε. Υπάρχουν προβλήματα συνεργασίας. Τώρα, για την αστυνομική αποστολή. Κύριε Κλάμπενχάουερ, πέστε μου συγκεκριμένα από την εμπειρία σας. Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να κάνουμε μετά το 2011. Είπατε ότι ενδεχομένως να μην ε, προχωρήσουν στην πάυση αυτής της αποστολής μετά το 2011. Μπορεί να μην σας κατάλαβα καλά. Ακόμα μια ερώτηση προς τον στρατηγό Μακόλ. Ως συντονιστής του ΝΑΤΟ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι τα γενικά σας συμπεράσματα για μια στρατή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάποια ερωτήματα και εγώ να θέσω. Ευχαριστώ τον στρατηγό, τον αρχηγό της, αστυνομι... τον αρχηγό της αστυνομικής αποστολής και τον κύριο Κλόπεν Χάουερ που είναι εδώ για να μας πληροφορήσουν πλήρως τι ακριβώς κάνουν. Κύριε Φέλερ, αναφερθήκατε στις επαφές που είχατε αναπτύξει με τις υπηρεσίες σας μεταξύ άλλων με το Μαυροβούνιο και άλλες χώρες οι οποίες επέτρεψαν να γίνουν κάποιες ενέργειες μεγάλης έκτασης για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και θα ήθελα γι' αυτό να θέσω το ερώτημα τι γίνεται στο στρατιωτικό αλλά και αστυνομικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τις επαφές με τη Σερβία, το Βελιγράδι δηλαδή, και με την Κροατία. Αυτό ξεπερνάει λιγάκι το το καθαρά στρατιωτικό και αστυνομικό θέμα, <clears throat> γιατί ασχολούμαι και με την πολιτική πτυχή. Ήμουνα πρόσφατα στο Ζάγκρεπ και μου είπαν ότι υπάρχουν ορισμένα προβλήματα που προκύπτουν από το γεγονός ότι κατά μεγάλη πιθανότητα οι Κροάτες στη Βοσνία Ζεχοβίνη θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις προεδρικές εκλογές της Κροατίας. Και κατά πάσα πιθανότητα εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να γίνει κάτι τέτοιο, αυτό θα μπορούσε να γύρει την πλάστικα υπέρ του ενός ή του άλλου υποψηφίου. Αυτό είναι θέμα λοιπόν ε, για την Κροατία. Υπάρχει το ερώτημα αν θα δοθούν σερβικά διαβατήρια στους πολίτες της Ρεπούμπλικας Σύρψκα. Όλα αυτά διατηρούν ζωντανή την πολιτική ένταση στην περιοχή και μου φαίνεται ότι δυσκολεύουν ή τουλάχιστον καθυστερούν την θεσμική εδραίωση και την πολιτική σταθεροποίηση. Γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν γέφυρες με άλλες όμορες χώρες. Πώς το βλέπετε λοιπόν το θέμα αυτό, είτε μέσα, στην, μέσα από την προοπτική των στρατιωτικών ή αστυνομικών σας δραστηριοτήτων, είτε σε ένα ευρύτερο πολιτικό επίπεδο. Ευχαριστώ κύριε Τα πιο σημαντικά ερωτήματα έχουν ήδη τεθεί. Θέλω να προσθέσω και το δικό μου ερώτημα. Πρώτα απ' όλα, δεδομένων των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η αμάλθεια από την αρχή και σε όλη την ύπαρξή της συνεργασίας με την Τουρκία επειδή δραστηριότητα Βερολίνου ΣΥΝ και το γεγονός ότι τώρα φοράτε δύο καπέλα. Εσείς έχει βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Στον ε, στρατηγό Φέλερ είπατε <clears throat> ότι πέρσι υπήρξε τέτραπλασιασμός των ε, ενεργειών ξεπλήματος χρήματος. Μπορείτε να μας ε, βοηθήσετε να, καταλάβουμε γιατί έγινε αυτό πέρσι. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά γιατί τετραπλασιασμός ιδιαίτερα πέρσι. Είχε να κάνει με την εσωτερική εξέλιξη της οικονομίας στη Βοσνία Ζεγοβίνη ή ήταν κάτι που είχε να κάνει με τον τρόπο με την οικονομική και χρηματοοικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε. Σας ευχαριστώ. Ε, Στατιέ Μακ Σας ευχαριστώ για τα ερωτήματά σας. Θα τις αντιμετωπίσω θεματικά και όχι κατά σειρά. Καταρχήν, το θέμα του μέλλοντος της αποστολής μας. Της εκτελεστικής μας ε, αποστολής. Εδώ η παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω είναι ότι η κρίση του αν είναι καιρός να περάσουμε σε άλλη, άλλο είδος αποστολής από μια εκτελεστική αποστολή εξαρτάται από το κατά πόσο αυτή η διαβρωτική και αντιπαραθετική πολιτική θα διευρυνθεί περισσότερο και σε άλλα πλαίσια. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, αλλά υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να γίνει αυτό στο μέλλον. Αυτή είναι μια πολιτική κρίση και μια κρίση στρατιωτικού χαρακτήρα. Εγώ από στρατιωτική έποψη θεωρώ ότι δεν υπάρχουν δείκτες αυτή τη στιγμή που δείχνουν ότι κινδυνεύει να υπάρξει μια κλιμάκωση σε στρατιωτικό επίπεδο. Ένα άλλο στοιχείο είναι η συνεκτικότητα της παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί είναι σημαντικό να παίξει ένα ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ερώτημα αν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει την αντιπαράθεση σε ρητορικό επίπεδο μεταξύ των εθνωτικών ομάδων. Εγώ νομίζω ότι όσο πιο πολύ κεντρική είναι η προσέγγιση μας, όσο πιο πολύ συνεκτική είναι η Ευρώπη με τη συνθήκη τη Λισαβόνα, τόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα. Γι' αυτό θέλουμε να εξασφαλίσουμε τη συνεκτικότητα ταχύτερα δυνατό. Επομένω, εγώ δεν αποκλίνω από την απόφαση αυτή αλλά φυσικά αυτή η απόφαση εξαρτάται από μία πολιτική αξιολόγηση για το αν μπορεί να υπάρξει έλεγχος αυτών των πολιτικών δυνάμεων στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Αυτό δεν είναι θέμα για ένα στρατιωτικό. Για το τώρα τι θα γινόταν αν εμείς τροποποιούσαμε την εντολή από μια εκτελεστική εντολή, <clears throat> αν χρειαζόταν λοιπόν να, να, και πάλι. Ναι, προφανώς θα χρειαζόταν μια νέα πολιτική εντολή. Αυτό είναι απαραίτητο. για τις πολιτικές κατευθύνσεις. Γνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες διαφωνίες σε σχέση με τη σωστή χρονική στιγμή. Αυτή τη στιγμή η αναθεώρηση θα φτάσει προς το τέλος του χρόνου. Έχουμε την απόσυρση στρατιωτών από το θέατρο επιχειρήσεων που μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Εγώ δεν θα ήθελα να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά δεν υπάρχει ακόμα συνένεση για την εκτελεστική εντολή. Αυτό το οποίο σημαίνει αυτό είναι ότι θα παραμείνουμε με ένα περιορισμένο αριθμό στρατιωτών επιτοπίως, κάτι το οποίο δυνητικά θα έχει επιπτώσεις. Και αυτό δεν είναι επιθυμητό, γιατί μπορεί να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου μπορεί να χρειαστεί να δραστηριοποιηθούμε σύντομα ή έχουμε <clears throat> κόδωνες κινδύνου και δεν θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε εγκαίρως τις εξελίξεις αυτές από στρατιωτική άποψη εγώ ανησυχώ γιατί μπορεί να μην μπορούμε να αντεπεξέλθουμε σε καταστάσεις οι οποίες θα δημιουργηθούν και να μην μπορούμε να βοηθήσουμε την κυβέρνηση της Βοσνίας Ερζεγοβίνη. Αν εσεί πιστεύετε ότι είναι σταθερή πολιτικά η κατάσταση και είσαστε έτοιμοι να δεχτείτε αυτό το κίνδυνο που είναι ένα πολιτικό κίνδυνο και όχι κίνδυνο ασφαλεία, εντάξει, τότε αυτή είναι μια απάντηση η οποία είναι πολιτικά αποδεκτή. Εγώ θα, απο, θα δώσω συνέχεια στο επίπεδο στο οποίο είμαι αρμόδιος. και θα πρέπει να προσαρμόσω το σχεδιασμό μου. Το επόμενο θέμα ήταν ο δικός χάρτης και η πρόοδος. Έχουν υπάρξει συμφωνίες καταρχήν, αλλά το ετήσιο σχέδιο το οποίο θα παρουσιαστεί το φθινόπωρο θα εξαρτηθεί και από την ε, επίλυση εσωτερικών θεμάτων σε ό,τι αφορά εγκαταστάσεις άμυνας. Και αυτό το θέμα πρέπει να επιληθεί εσωτερικά. Υπήρξαν μεγάλες διασκολίες για να υπάρξει συμφωνία μέχρι στιγμής. Για την αποστολή κατάρτισης. Η συμφωνία να προχωρήσει αυτή η αποστολή ελήφθη τον ε, Ιανουάριο και έχουμε δημιουργήσει ένα τέτοιο μηχανισμό που θα μας επιτρέψει να προωθήσουμε αυτή την ε, διαδικασία με ομάδες που έρχονται από τα κράτη-μέλη για να υπάρξει σωστή κατάρτιση Στι αναπλές δυνάμει της Βοσνίας Ερζεγοβίνη και να υπάρχει μεγαλύτερη συνεκτικότητα. Αυτό έχει τύχει ευρέω συντονισμού με το ΝΑΤΟ, γιατί και το ΝΑΤΟ συμβάλλει ιδιαίτερα στην ανάπτυξη τη αμυντική ικανότητα κτλ. Ε, μαζί με Υπουργεία Αμυνα και Υπουργεία Οικονομικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται περισσότερο στο τακτικό επίπεδο και έχουμε κάνει μια σημαντική συμβολή στον τομέα αυτό για το σχεδιασμό των ενεργειών κατάτησης και εμείς θα πράξουμε εξάλλου κάτι τέτοιο και στο Αφγανιστάν. Η σχέση μας λοιπόν στον τομέα αυτό εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ θετική. Η σχέση μας με τους δικαστές είναι πολύ θετική και ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο στο οποίο οι τοπικές αρχές θα πρέπει να αναλάβουν άμεση ευθύνη και όχι εμείς για τα όπλα τα οποία βρίσκονται στην Ήπεθρο. Υπάρχουν όπλα στην Ήπεθρο η πλειοψηφία τους κατέχονται από ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας. Εμείς τις παρακολουθούμε, η αστυνομία τις παρακολουθεί και σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των ε, πυροβόλων όπλων ε, που κατέχεται από ιδιώτες, αυτό είναι θέμα δικαίου, είναι θέμα νόμου και είναι θέμα επομένω της αστυνομία και όχι θέμα στρατιωτικής παρέμβαση. Πρέπει να καταφύγουμε στρατιωτική παρέμβαση μόνο στο τέλος, όταν έχουν εξαντληθεί όλες οι άλλες οδοί. Σε ό,τι αφορά ε, της για την Τουρκία. Δεν καταλαβαίνω τα σχόλια. Ε, εγώ στρατιωτικός μπορώ να πω ότι η Τουρκία είναι απόλυτα επαγγελματική, πολύ αποτελεσματική και μας βοηθάει τα μάλα. Ε, και ποτέ επί τόπου ε, δεν κατάλαβα ή αντελήφθη διάφορες δυσκολίες μεταξύ των επαφών που έχει η Τουρκία με τον τοπικό πληθυσμό. Νομίζω ότι χρησιμοποιείται θετικά και, εγώ θα πρέπει να, και εμείς θα πρέπει να ενθα, ενθαρρύνουμε την βοήθεια από την Τουρκία. Τα μαθήματα τώρα από το Βερολίνο Plus ε, μας δείχνουν ότι μπορούν να γίνουν πάρα πολλά όταν το Ευρωπαϊκό, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ συνομιλούν. Μπορούν να συνομιλήσουν για ένα θέμα και πρέπει να μιλήσουν για ένα θέμα, το οποίο ποιο είναι η Βοσνία-Ζεγοβίνη η στατιωτική επιτροπή του ΝΑΤΟ και η στατιωτική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούν και συζητάνε ένα θέμα, μόνο τη Βοσνία. Εγώ βλέπω τι μπορεί να γίνει στη Βοσνία. Όταν ε, βλέπετε ότι οι λύσεις ε, γενικά στο, στα προβλήματα της Βοσνίας αφορούν την πολιτική και την οικονομία, η συνεισφορά του στρατού είναι πολύ συγκεκριμένη, πολύ εστιασμένη. Αν εμεί δεν τα καταφέρουμε, θα χαθούν ζωέ πολιτών και θα χαθούν ζωέ στρατιωτικών. Επομένω, πρέπει να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, στρατηγέ μου, ο κύριο Κλάν Πενχάουερ. Θα ήθελα να επαναλάβω κι εγώ. Τα δέχομαι αυτά που άκουσα, τα περισσότερα από αυτά που είπε ο στρατηγός για τη συνεργασία ΝΑΤΟ και Ένωση στη Βοσνία. Ένα ευρύτερο θέμα όμως υπάρχει για την μετάβαση και την προενταξιακή διαδικασία. Δύο πτυχές έχει αυτό το πρόβλημα. Πρώτον, Αυτή τη στιγμή καθορίζουμε πρότυπα και benchmarks για να μπορέσουμε να λάβουμε μια απόφαση. Και θέλουμε να συνδυάσουμε τα αποτελέσματα για να δούμε αν είμαστε σε θέση να μιλήσουμε για ένταξη. Το δεύτερο θέμα είναι ο παράγοντας της όθησης, push factor. Μην ξεχνάτε ότι ο πολιτικός εξτρεμισμός είναι κάτι που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα χώρο να μειώσουμε την ατιμορρησία, να καταστεί επικίνδυνο να θέλει κάποιος να καταχραστεί την εμπιστοσύνη των άλλων. Um, um, Ο κύριος Φέλε προσπαθεί και αυτός με τους συναδέλφους του της αστυνομίας να δημιουργήσει μια συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αστυνομικών οντοτήτων που υπάρχουν και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι έτσι ξεπερνιούνται οι ψυχολογικοί φραγμοί που ακόμη υπάρχουν. Πρέπει να μάθουν όλοι να συνεργάζονται. Γι' αυτό και οι μεγάλες εθνικές επιχειρήσεις καταπολέμησης του εγκλήματος είναι κάτι που είναι πολύ καλό παράδειγμα για συνεργασία. Καμιά φορά τα αναλαμβάνει η Ομοσπονδιακή Αστυνομία, καμιά φορά η αστυνομία της Ρεπούμπλικας Σούρπσκας. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες κάποιας βιωσιμότητας και αυτό θα είναι το τελικό κριτήριο. αν δηλαδή υπάρχει αυτή η βιωσιμότητα για να επιτρέψει την ένταξη. Είναι βέβαια σωστό ότι οι πολιτικές επιχειρήσεις είναι λιγότερο ακριβές από τις στρατιωτικές, αλλά και αυτές κάποτε πρέπει να περάσουν στους τοπικούς παράγοντες. Και νομίζω ότι θεμητό θα ήταν να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πότε θα γίνει η μεταβίβαση αυτών των δικαιοδοσιών πλήρως στους τοπικούς. Ο κύριος Φέλλερ. Ευχαριστώ πολύ. Περίπου τα ίδια έχω, θα είχα και εγώ να πω, όχι ακριβώς τα ίδια. Πιστεύουμε ότι μετά το 2011 θα αρχίσει να τίθεται αυτό το θέμα της πολιτικής απόφασης και εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να χορηγούμε την πολιτική συμβουλή που χρειάζεται για να ληφθεί αυτή η απόφαση. Υπενθυμίζω ότι, ότι ακόμη είμαστε σε μια προσπάθεια οικοδόμησης όχι μόνο εμπιστοσύνης αλλά και θεσμών. και είδαμε ότι έχουν υπάρξει προσπάθειες απλοποίησης και καλύτερης οργάνωσης των διαδικασιών δίωξης του οργανωμένου εγκλήματος. Και με τα δύο νομοσχέδια αστυνομικής μεταρρύθμισης την άνοιξη του 2008, μετά από τα νομοσχέδια αυτά, άρχισε να εφαρμόζεται και ένας συντονισμός των αστυνομιών. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμη 17 διαφορετικές οντότητες σε ομοσπονδιακό, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο. 17, εγώ χρειάζομαι πολλές φορές να συνομιλώ με 17 τοπικούς παράγοντες. Χρειάζεται λοιπόν κάποια απλοποίηση και αυτό ισχύει για όλους τους παράγοντες και για το ανώτατο κρατικό επίπεδο. Πολλοί έχουν την πολιτική θέληση να μπορέσει και σε ομοσπονδιακό επίπεδο να υπάρξει μία ένα συντονισμό των δραστηριοτήτων δίωξης του κλίματος όπως γίνεται σε τοπικό επίπεδο. Εμείς όμως δεν βασιζόμαστε σε εντολή βάση του κεφαλαίου 7 και αν και για να ληφθεί οποιαδήποτε πολιτική απόφαση για την, ενταξιακό, την ενταξιακή πρόπτικη θα πρέπει να μην ξεχνάει ότι εμείς εκλήθημεν από την Προεδρία της Βοσνίας Ρεγοβίνης να έρθουμε και ότι όσο κρατάει η εντολή μας Θέλουμε να ενδυναμώσουμε θεσμικές διαδικασίες στον τομέα του συντονισμού, της συνεργασίας και της επικοινωνίας. Αυτό ακριβώς πρέπει να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε και είναι επιτυχία ότι οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες και οι αστυνομικοί καταφέραμε να καταλήξουν σε κάποια συνεργασία και συντονισμό, θεσμικά εννοώ, και σε κρατικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό είναι εξαιρετική εξέλιξη. Σε τεχνικό επίπεδο το Ζάγκρεμπ, το Βελιγράδι ή οποιαδήποτε άλλη πόλη δεν έχει πια πρόβλημα επικοινωνίας με τους υπόλοιπους για θέματα δίωξης εγκλήματος. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι τους τελευταίους μήνες ε, έχουν χειροτερέψει λίγο τα πράγματα, αλλά αυτό είναι πολιτική κρίση και δεν θα την κάνω εγώ. Η δυνατότητα συνεργασίας σε νομικά θέματα πρέπει κάποτε βέβαια να αναλυφθεί από τους τοπικούς παράγοντες και είναι από τα σημαντικότερα από τους σημαντικότερους στόχους μας να υπάρξει δηλαδή αυξημένη τοπική δυνατότητα ανάληψης αυτών των καθηκόντων. Όταν θα χρειαστεί να αποφασιστεί η ενταξιακή προοπτική, θα χρειαστεί να αξιολογήσουμε και εμείς το ότι οι εκλογές του Οκτωβρίου 2010 θα μας δείξουν πού βρισκόμαστε ως προς την πολιτική δυνατότητα του συστήματος της Βοσνίας Ερζεγοβίνης να αντιδράσει καταλήλως. Γιατί η ένομη τάξη δεν μπορεί να διαχωριστεί από, από το υπουργικό επίπεδο και Υπάρχει μεν τεχνική πρόοδος, αλλά πρέπει να δούμε αν υπάρχει και πολιτική. Από συνομιλίες που είχαμε υπουργούς, στους οποίους θέλησα να δείξω ότι όλα αυτά πρέπει να μεταφραστούν και σε πολιτικό επίπεδο διαδικασίας λήψης αποφάσεων, είδα ότι κατανοούν οι περισσότεροι ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο. Για το ρόλο της Τουρκίας έχουμε τρεις αστυνομικούς και δύο μη αστυνομικού στην αποστολή μας οι οποίοι είναι πολύ καλοί είναι πραγματικοί εμπειρογνώμονες δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα λύνουν προβλήματα λύνουν οι Τούρκοι και έχω συνεργαστεί και άλλες φορές με εγκληματολόγους Τούρκους και ξέρω ότι η συνεργασία μαζί τους είναι πολύ καλή Τέλος αυτά που είπε η κυρία Γκόμες για, την, ε, για το ξέπλυμα βρωμίκου χρήματος. Υπάρχει αυξανόμενη καχυποψία για τις χρηματικές δοσοληψίες και αυτό δείχνει ότι το σύστημα είναι διατεθειμένο να καταπολεμήσει το ξέπλυμα αυτό και να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα σοβαρά. Ο Υπουργός Ασφαλείας μας κάλεσε να δώσουμε και εμείς συμβουλές για τον καλύτερο δυνατό τρόπο λειτουργίας του τμήματος ε, χρηματικών πληροφοριών ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει διάθεση ειλικρινής από τους τοπικούς εθνικούς παράγοντες. Και εμείς θέλουμε απλώς να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα εξαρτάται από πρόσωπα αλλά από θεσμικές διαδικασίες. Αυτό θα κάνουμε το επόμενο, επόμενο 1,5 χρόνο. Ευχαριστώ κύριε, κύριε Χάουερ. Ευχαριστούμε κύριε στρατηγέ μας για την πολύ σαφή παρουσίαση της ε, αποστολής σας. Εγώ δεν γνωρίζω πολύ καλά την ε, Συμφωνία Βερολίνου ΣΥΝ. Με ενδιαφέρει όμως ιδιαίτερα το πώς αλληλεπιδρούν οι δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, αν υπάρχουν εθνικές επικαλύψεις και συγκρούσεις και καταλαβαίνω ότι το Βερολίνο ΣΥΝ το αντιμετωπίζει αυτό κατευθείαν. Αυτό θα ήθελα να ξέρω αν υπάρχει σπατάλη προσπαθειών και επικάλυψη προσπαθειών, μήπως έχετε πάρα πολλούς οι οποίοι παίζουν συγχρόνως στο γήπεδο της Βοσνίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπούτικ Όφερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε την δυνατότητα να ρωτήσω και πάλι. Σίγουρα είμαι σκεπτικιστής σε ό,τι αφορά τις ελπίδες που τρέφουν ορισμένοι. Είμαι σκεπτικιστής εναντί της δυνατότητας να υπερπηδηθούν οι πολιτικές δυσκολίες σε απόλυτο επίπεδο και να μην έχουν επιπτώσει στον τομέα της ασφάλειας. Εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει μια αξιόπιστη παρουσία ασφάλεια στην Βοσνία Ζεχοβίνη, αλλά φαίνεται ότι η πολιτική αστάθεια στην ε, Βοσνία Ζεχοβίνη δεν επιτρέπει να εξασφαλιστεί αυτή η ασφάλεια. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω και πάλι με αυτή την ευκαιρία για το ρόλο της Προεδρίας στην Βοσνία Ζεχοβίν, Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι από την πλευρά της Προεδρίας στη Βοσνία Ζεχοβίνη η συνέχιση της παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επιθυμητή και πώς ακριβώς θα μπορούσε η παρουσία των κατών μελών που εμπλέκονται στην Αλθέα να υπάρξει μια μεγαλύτερη συμμετοχή των εκπροσώπων της Προεδρίας της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Σε ποιο βαθμό υπάρχουν λοιπόν τακτικές επαφές με τον πρόεδρο της Βοσνίας Ερζεγοβίνης για να μιλήσουν για το μέλλον της Αλδίας. Ή εμείς απλώς ε, αποφασίζουμε χωρίς να λάβουμε υπόψη της την απόψη της Προεδρίας της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Ο στρατηγός Μακ Κάου Μεσή, ο στρατηγό. Βερολίνο ΣΥΝ. Οι ρυθμίσει του Βερολίνο ΣΥΝ είναι περιπτώσει όπου το ΝΑΤΟ λειτουργεί σε στρατιωτικό επίπεδο και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολιτικό επίπεδο και επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ των δύο. Αμφωτέρων και των δύο δηλαδή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί έτσι να επωφεληθεί από την δομή διοίκηση του ΝΑΤΟ και τη δομή επι Μελητεία και αυτό επιτρέπει να υπάρχει διάλογο, συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών. Κατά την άποψή μου υπήρξε πολύ επωφελή αυτή η διαδικασία και αποτελεσματική του Βερολίνου ΣΥΝ και στου δύσκολου αυτού καιρού, όπου όλοι θέλουν να εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα είναι ένα πολύ καλό τρόπο να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο του πόρου που υπάρχουν. Από την άποψη αυτή και βάσει τη δική μου εμπειρία. είναι πολύ αποτελεσματικός τρόπος να λειτουργήσουμε σε ό,τι αφορά τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ σε άλλα θέατρα. Εκεί που έχουμε την μεγαλύτερη επίδραση είναι το Αφγανιστάν με την ISAF και την UPOL και φυσικά η ULEX και η EU4 στην πρώην Ιουκοσλαβία. Επίσης και στην ανοιχτή θάλασσα στα πλαίσια της Αταλάντης. Το πλαίσιο το οποίο έχει δημιουργηθεί βέβαια τυπικά, δυσκολεύει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο δύναμεων. Και άκουσα αυτά που είπε ο κ. Κάμπελ για τη θαυμάσια συνεργασία που γίνεται στην περίπτωση της ΚΕΙΦΟΡ. Είναι θαυμάσια συνεργασία, αλλά θα πρέπει να είμαστε σαφεί ότι είναι άτυπη αυτή η συνεργασία, είναι τακτικού χαρακτήρα. Και το λέω αυτό με κάποιου δισταγμού, αλλά αλλά πρέπει να πω ότι μερικές φορές η συνεργασία γίνεται σε πείσμα των πολιτικών ρυθμίσεων. Είναι μια παράξενη κατάσταση όπου πρέπει να βασιζόμαστε στους στρατιωτικούς να κάνουν κάτι το οποίο δεν είναι αυτό που τους έχουν πει να κάνουν. Αυτό εμποδίζει λοιπόν και μια συνολική αντιμετώπιση. Ξέρουμε σε πάρα πολλέ επιχειρήσεις ότι η διακυβέρνηση και η επίτευξη των σωστών στόχων εξαρτώνται από την αναγνώριση όλων των πλευρών ότι υπάρχει κοινό συμφέρον. Λοιπόν, ο διάλογος μεταξύ των δύο φορέων πρέπει να συμβάλλει σε μεγαλύτερη σαφήνεια και διευκρίνηση των προβλημάτων. επιτοπιως βλεπετε βλέπετε ότι υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ U4 και, K, και ULEX, μεταξύ ISAF και UPOL κτλ. Αλλά δεν θα έπρεπε να είναι υποχρεωμένη να τα κάνουν αυτά εκτός πλαισίου. Θα πρέπει να έχουν ένα πλαίσιο το οποίο αντί να δυσκολεύει τα πράγματα θα πρέπει να του βοηθάει και δεν πρέπει να τους επιτρέπει και να τους αναγκάζει να κάνουν άτυπα δίκτυα <clears throat> επικοινωνίες. Αυτό είναι πραγματικά ένα πολιτικό πρόβλημα το οποίο μας βάζει μας σε μια πολύ δύσκολη θέση. Ευχαριστώ πολύ. Για την άλλη ερώτηση που κάνατε, αν κατάλαβα καλά. Την άποψη της Προεδρίας Βοσνίας Ερζεγοβίνης ε, για την Αλθέα. Αυτό είναι ευαίσθητο και πολιτικό θέμα και το αφήνω στους πολιτικούς, αν δεν σας ε, πειράζει. Για την ε, συνεργασία με την Αλθέα Συνεργαζόμαστε με τους πολιτικούς. Μας βοηθούν και η συνεργασία αυτή είναι πραγματικά παραγωγική. Το μόνο που μπορώ να πω είναι αυτό. Euh, ευχαριστώ το στρατηγό. Ο ταξίρχος Φέλερ, μήπως θα ήθελε να κάνει κάποιο σχόλιο. Όχι. Καλύφθηκαν όλα τα θέματα. Σας ευχαριστώ και τους τρεις. Θα σας ξαναδούμε στην ακρόαση που θα κάνουμε για το ΝΑΤΟ. Μετά από την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ που έγινε στη Ρήγα και την ημέρα που είχαμε χθε, θα θέλαμε να ξανασυζητήσουμε την αναθεώρηση της στρατηγικής συγγνώμη, αντίληψης του ΝΑΤΟ. Θα κάνουμε μια συζήτηση για τις ε, απόψεις του ΝΑΤΟ για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τα ξαναπούμε στις 23 Ιουνίου για την επόμενη συνεδρίασή μας. 23 Ιουνίου η επόμενη συνεδρίασή μας. Γεια σας και ευχαριστώ.